Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σα. Καλημέρα σα, κύριε Γκάλερ. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η ψηφοφορία για την έκθεση σχετική με την κατάσταση στο Αυγαριστάν έχει αναβληθεί. Άλλε ανακοινώσει δεν έχω, για τα πρακτικά έχετε τίποτα. Όχι. Εγκρίνει τη μυρίσια διάταξη. Σημείο 4. Καλωσορίζω τον κύριο Πέτερ Μάουρερ, πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσατε να διαθέσετε το χρόνο για να έρθετε σε εμάς σήμερα. Γιατί νομίζω ότι είναι αναρρύθμιτος να ρίχνετε τα προβλήματα που χρειάζεται ανθρωπιστική υποστήριξη από την Ουκρανία με τόσους πολλούς ε, εκτοπιστέντες. Το Ιράκ, τη Συρία, την Ιεμένη, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, θα μας απασχολήσει και πιο μετά, Νότιο Σουδάν και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου που έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα και ροές προσφύγων. Αυτά που λέμε και ευρύτερη γειτονία, αλλά όχι μόνο. Είναι οι περιοχές που δραστηριοποιήσετε. Πάντα έχετε πολύ καλή συνεργασία με την Ερυθρά Εμισέλινου. Πολύ ικανοποιητική συνεργασία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζει. Σας διαβεβαιούμε ότι έχετε όλοι μας την υποστήριξη. Θέλουμε πάνω απ' όλα όμως να ακούσουμε τι έχετε εσεί να πείτε. πώ κρίνετε την κατάσταση και τι είδου συγκεκριμένε προτάσεις μπορείτε να μας κάνετε για να βοηθήσουμε και εμεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχετε τον λόγο. Κύριε Μάουρερ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε και κύριοι, Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να είμαστε εδώ μαζί σα σήμερα και να σας ενημερώσω για τις ε, βασικές ανησυχίε ε, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, της Διεθνή Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και το τι ακριβώς κάνουμε. Καταρχάς, ε, εισαγωγικά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να σας πω ότι το σημαντικότερο ζήτημα τα τελευταία χρόνια είναι ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων δυνάμεων είτε σε παγκόσμιο είτε σε περιφερειακό επίπεδο κάτι το οποίο προσφέρει ένα περιθώριο για διάφορες μορφές στρατιωτικών και ένοπλων λύσεων, διάφορες ομάδες αναζητούν ε, να καταλάβουν διάφορες περιοχές ε, ε, στην ευρύτερη περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ούτε κάποια ομάδα χωρών έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή να επιβάλλει την τάξη και ένα διεθνές σύστημα το οποίο θα ε, επιφέρει πολιτικές λύσεις σε όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις ε, στις οποίες δραστηριοποιούμεθα. Ως ε, ανθρωπιστική οργάνωση λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον της εξής κατάστασης. Τα τελευταία τρία χρόνια υπήρχαν ε, ε, συνεχώς νέες ε, σειράξεις σε μηνία βάση σχεδόν και έχουμε θύματα εκτοπισμένους, εσωτερικώς εκτοπισμένους και πρόσφυγες. θα έχετε διαπιστώσει ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε πλέον το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων και μέχρι σήμερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό εσωτερικώς εκτοπισμένων. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατεύθυνση. Ο αριθμός και ε, η σοβαρότητα των συγκρούσεων είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ σημαντικές προκλήσεις, αλλά Επίσης είναι το γεγονός ότι οι σειράξεις αυτές προσλαμβάνουν όλο και περισσότερο περιφερειακή διάσταση. Πριν από τρία χρόνια αναφερόμασταν στη ε, σύγκρουση της Συρίας, σήμερα αναφερόμαστε στη Μέση Ανατολή και ε, είναι όλη η περιοχή μπλεγμένη. Επίσης ε, αναφερόμασταν πριν από τρία χρόνια στην κρίση στο Μάλι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η κρίση στο Σαχέλ και πρόκειται για μια ε, περιοχή μεταξύ Λιβύης και ε, Βόρειας Νιγηρίας. Πριν από κανένα δύο χρόνια αναφερόμασταν στη Σομαλία ή στο Σουδάν, αλλά αυτή τη στιγμή πρόκειται για περιφερειακή κρίση. Έχουμε και την Αιθιοπία η οποία έχει βρεθεί εν μέσω και ε, φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στην Αφρικανική Ήπειρο. Επομένως, οι κρίσεις δεν είναι μόνο περισσότερες σε αριθμό, αλλά είναι και περιφερειακές και πρέπει να προσθέσω ότι είναι και συστημικές, που σημαίνει ότι ως ε, άνθρωποι που ασχολούμαστε με τις ανθρωπιστικές λύσεις ε, δεν έχουμε απλώς να ανταποκριθούμε σε βραχυπρόθεσμες ανάγκες σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον συμμετέχουμε σε ε, μεγαλύτερες παρατετημένες ε, συστημικές σειράξεις. Και τι εννοώ με τον όρο συστημικός. αν δούμε τι γίνεται στη Συρία και στη Λιβύη, σημαίνει ότι καταραίουν τα συστήματα υγείας, το, τα συστήματα υδάτων, ε, το υγειονομικό σύστημα. Υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι σε περιοχές που δεν έχει νερό και υπάρχει νερό εκεί που δεν έχει ανθρώπους. αυτό συμβαίνει λόγω των εκτοπισμών που έχουν προκύψει από τις σειράξεις. Κατοικίες, υγεία, υγειονομικά συστήματα, νερό, σχολεία, όλα αυτά καταραίουν. Μόλις ήρθα από τη Βορεια Ανιγυρία, ήμουν στο Μαντκούρ την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί έκλεισαν σχολεία και κλείνουν σχολεία τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Δεν πάει σχολείο κανένα παιδί εδώ και δυόμιση χρόνια, εκτός από τα Ισλαμικά σχολεία. Είναι ιδιωτικά και αυτά είναι ακόμα ανοιχτά. Αλλά τα δημόσια σχολεία δεν ε, ε, λειτουργούν. Αυτό είναι λοιπόν η παρατηρήσή μου. Δεν έχουμε απλώς μια προσωρινή ε, μετακίνηση κάποιων ανθρώπων. Ε, ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό σειράξεων, δεν είχαμε τόσο μεγάλες ε, και βαθιές σειράξεις και δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη κατάρρευση συστημάτων. Ε, πλέον βρισκόμαστε λοιπόν στο ζενήθ και νομίζω ότι δυστυχώς το σύστημα ανταπόκρισης της διεθνούς κοινότητας δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Έχουμε συνεχώς ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ των αναγκών που είναι εκθετικά αυξανόμενες και ε, των δυνατοτήτων που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Και όταν λέω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά θα ήθελα να προσθέσω και το εξής ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ε, όλο ένα και περισσότερο νιώθει απόλυτα μόνος σε διάφορες περιοχές ε, σειράξεων ανά τον κόσμο, διότι δεν ε, υπάρχει κανείς άλλος για να έρθει σε κάποιες από τις χειρότερες περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Αφγανιστάν, Νότια Σομαλία, Λούγκανς και Κεντόνιες, ε, η λίμνη του Τσάντ, ε, η Ονίγυρα, η Νιγηρία, Βόρειο Μάλι. Αυτές είναι περιοχές τις οποίες η Επιτροπή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ε, και κάποιες άλλες ε, επιτροπές και οργανισμοί του, Διεθνούς, ε, του Ερυθρού Σταυρού που έχουν κάποιες δομές είναι οι μόνες δομές που υπάρχουν επιτόπου σε αυτές τις περιοχές. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία θα ήθελα να σας θέσω ως πολιτική και ε, υπάρχει το γεγονό ότι ο κύριος Μπροκ ε, μου ζήτησε να κάνω κάποιες προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε κατά πόσον η χρηματοδότηση που επιλέγεται χρησιμοποιείται με κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις προτεραιότητες που έχουμε σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Και νομίζω ότι θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των αναγκών που αναλύεται και των ροών χρημάτων και το προς τα που διοχετεύονται αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξανασκεφτεί την ισορροπία μεταξύ ανθρωπιστικής συνδρομής και αναπτυξιακής βοήθειας. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες σήμερα προκειμένου να εγγράψουμε τις δράσεις μας στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των, ε, κοινωνιών, διότι πλέον είναι ε, πολύ μεγαλύτερο το διάστημα στο οποίο συμμετέχουμε σε αυτές τις δραστηριότητες, αλλά θα πρέπει να καθορίσουμε και σωστά τους στόχους μας και εκεί έρχεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς συμμετέχουμε σε κάποιες από τις σοβαρέτερες κρίσεις και εκεί διαπιστώνουμε ότι έχουμε ελάχιστους, αν όχι και κανέναν, από πλευράς αναπτυξιακής. Ε, το ερώτημα είναι λοιπόν κατά πόσον οι πόροι διοχετεύονται στη σωστή κατεύθυνση, κατά πόσον δαπανώνται ε, ώστε να σταθεροποιούν, ή να βοηθούν στη σταθεροποίηση των πιο ευάλωτων περιοχών ή όχι. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι το εξής. οι, διεθνεί διεθνείς οργανισμοί, η Παγκόσμια Τράπεζα, η ε, Παγκόσμια Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι κατάλληλα εξεπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ευάλωτες καταστάσεις που διαπιστώνουμε στις περισσότερες σειράξεις σήμερα. Και επίσης να σας πω και τι με ανησυχεί. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι όλο ένα και περισσότερο βρισκόμαστε σε ε, περιπτώσεις που υπάρχουν ευάλωτες καταστάσεις και καταστάσεις σύγκρουσης σε χώρες μεσαίου εισοδήματος. Και χώρες μεσαίου εισοδήματος δεν ε, είναι επιλέξιμες για να πάρουν αναπτυξιακή βοήθεια από τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Ε, Παραδείγματο χάρη, η Ουκρανία δεν είναι φτωχή χώρα, αλλά εν τέλει ο ε, Ερυθρό Σταυρό είναι ο μόνος ο οποίος δίνει ανθρωπιστική βοήθεια εκτός από τα ρωσικά κομβόη που έχουμε στις ε, πόλεις του Ντόνετσκ. Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, αυτές είναι χώρες μεσαίου δήματο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν να λάβουν αναπτυξιακή βοήθεια για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν και να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες αυτής της κρίσης και δεν ξέρω κατά πόσον η διεθνή κοινότητα είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τρίτον, μπορεί να είναι λίγο φτηνό το επιχείρημά μου, αλλά ως άνθρωπος που είμαι ανθρωπιστής, ε, ασχολούμαι με ανθρωπιστικά ζητήματα, κάθε μέρα με εκπλήσει το γεγονός ότι Υπάρχει ελάχιστος χρόνος και προσπάθεια που αφιερώνονται για διπλωματικές λύσεις ε, σειράξεων. Αυτό δεν είναι θέμα των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Εμείς προσπαθούμε να κρατηθούμε μακριά από αυτό. Αλλά είναι πολιτικό καθήκον και νομίζω ότι ως πολιτικοί, ως βουλευτές, ως άνθρωποι που, ασχολεί, ε, που ε, ασχολείστε με την εκτελεστική εξουσία σε κυβερνήσεις, ως μέλη των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ο κόσμος περιμένει διακαώς να υπάρξει μια δραστήρια διπλωματία η οποία θα ε, αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι εμείς ε, είμαστε εκεί για να προσφέρουμε ουδέτερη, αμερόληπτη βοήθεια και αν μπορούμε να την κάνουμε ξεχωριστά από τους πολιτικούς είναι ότι καλύτερο. Αλλά οι πολιτικοί και τα διάφορα πολιτικά βήματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε μέτρα μετριασμού των συναπιών χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις πηγές των προβλημάτων. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Ε, όταν ήμουν στο γραφείο του κυρίου Μπροκ, του ανέφερα ότι αυτή τη στιγμή η μετανάστευση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Εμείς τα τελευταία ένα-δύο χρόνια είχαμε ε, κάποιες εμπειρίες για το μετρασμό των ανθρωπιστικών κρίσεων ε, στις διάφορες μεταναστευτικές οδούς, στην Βόρεια Αμερική υπάρχουν ε, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Μισοέλληνο κάποιοι σταθμοί ε, τους οποίους ε, ε, στήσαμε ακριβώς για να βοηθήσουμε με τις επιστροφές και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κινούνται προς τα βόρεια. Αυτό δεν επιλύει βέβαια τα θέματα της μετανάστευσης, αλλά εμείς δεσμευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε <clears throat> στη Μεσόγειο ιδίως να κινητοποιήσουμε τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά η Στο Σαν Μαρίνο γίνεται τώρα μια συνάντηση των τοπικών ε, φορέων του Ερθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μισελίνου είναι απαραίτητο να δούμε αν μπορούμε σε ανθρωπιστικό επίπεδο να εργαστούμε για να μετριάσουμε κάποιο από τον αρνητικό αντίκτυπο που δημιουργείται στη Μεσόγειο από το πρόβλημα αυτό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις είναι το εξής. Θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και τα θύματα της βίας και ενάντια σε αυτούς οι οποίοι ασκούν βία. Όταν ήμουνα στην, στα προάστια της Δαμασκού, όταν ήμουνα στις γειτονικές χώρες της Συρίας και πάλι η δική μας δραστηριότητα, όσο δύσκολη και να είναι, βοηθάει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν είτε μέσα στη χώρα τους ή από τη χώρα τους, ενδεχομένως να έχουν περάσει σύνορα, μπορούμε τουλάχιστον ή δυνατόν να τους πείσουμε να μείνουν στην περιοχή αυτή. Εφόσον μπορούμε να τους δώσουμε με λογικό τρόπο ανθρωπιστική βοήθεια για να παραμείνουν κοντά στις ευθείες τους. Ήθελα λοιπόν να κάνω αυτές τις λίγες παρατηρήσεις και να σας αναφέρω τις σκέψεις αυτές και πάντα ενδιαφέρομαι να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις <clears throat> και να απαντήσω ή μπορώ στα δικά σας ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος Μπλοκ. Ο κύριος Βαϊράνεν, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΕΒΑ. Κάνουμε μια κοινή συζήτηση με την Επιτροπή ΔΕΒΕ Ανάπτυξης, όπως ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάουρερ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Πιστεύω ότι ως Επιτροπή Ανάπτυξης εμείς οπωσδήποτε χαιρετίζουμε τις ε, επιθυμίες που διατυπώσατε για το μέλλον. Ήθελα και εγώ να κάνω μια μικρή προσωπική συμβολή στα, στην προβληματισμό για τα θέματα αυτά και έχω διανύμει ένα άρθρο σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της υπάτης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αλλά φυσικά και την οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού. Διάβασα στους χθεσινούς Financial Times για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Λιβύη, στα κέντρα κράτησης. Αναφέρθηκε και το θέμα του Ερυθρού Σταυρού, συγκεκριμένα. Δεν έχουν γίνει λοιπόν αρκετά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δυσχερή συνθήκε σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κέντρα για υποδοχή προσφύγων στη νότια όχθη της Μεσογείου, ώστε αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν εκεί. Ίσως και οι πρόσφυγες από τη Λιβύη μπορούν να μπουν σε αυτούς τους καταβλισμούς αντί να μένουν σε φυλακές στη Λιβύη. Αν μπορέσουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια τέτοια ανθρωπιστική λύση, αυτό θα μας επιτρέψει να ελέγχουμε καλύτερα τα βόρεια τη βόρεια ακτή της ε, Αφρικής και να μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτούς που προσπαθούν παράνομα να έρθουν στην Ευρώπη και να τους κρατούμε σε αυτά τα κέντρα <clears throat> προσφύγων όπου η πάτη αρμοστία μπορεί πράγματι να διακριβώνει ποιοι από αυτούς έχουν το δικαίωμα ασύλου και επομένως τα κρατημέλη μέσα στα πλαίσια των εθνικών ποσοστώσεων μπορούν να τους υποδέχονται στο εδάφο του. Πιστεύω ότι η ιδέα του να έχουμε υποχρεωτικέ ποσοστώσεις για τους ετούντε ασύλου που είναι ήδη στην Ευρώπη, αυτό δεν είναι μια καλή ιδέα. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρξει μια ποσόστοση σε συνάρτηση με το σύστημα της υπάτης ε, αρμοστίας του ΟΗΕ και να παίρνουμε πρόσφυγες από τους καταβλισμούς της υπάτης αρμοστίας. Ε, ελπίζω θα μπορέσετε να διαβάσετε το σημείωμα μου. Έχω δώσει και ένα αντίγραφο στον κύριο Μάουρ. Ελπίζω ότι μπορείτε να το υποστηρίξετε. Σε σχέση με το έργο τώρα της Επιτροπής Ανάπτυξης, θέλω απλώς να πω ότι αντιμετωπίζουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και τα ανθρωπιστικά θέματα. Ο συνδυασμός των δύο θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα, εστιάζουμε περισσότερο στην προετοιμασία για την πρώτη που έχει γίνει ποτέ διάσκεψη κορυφής για τα ανθρωπιστικά θέματα, όπως ζήτησε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Θα γίνει αυτή η διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη το Μάιο του 2016. Ο στόχος θα είναι να προσαρμόσει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Σύστημα στο αναδυόμενο στερέωμα καταστάσεων εκτάκτης, εκτάκτου ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η ανθρωπιστική βοήθεια οι προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μισελίνου συνάδουν ιδιαίτερα με τις ευρωπαϊκές αρχές της αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και οικουμενικότητας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Προετοιμάζοντα λοιπόν αυτή τη διάσκεψη κορυφή τη Κωνσταντινούπολη, η Επιτροπή μου θα προσπαθήσει να ενισχύσει τι προσπάθειε για ένα αποτέλεσμα που θα είναι θετικό και θα καθοδηγείται από αυτέ τι αρχέ προ όφελο των δικαιούχων. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Μάουρερ για την θαυμάσια ε, παρουσίασή σας και τώρα φυσικά θα περάσουμε στις ερωτήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, καθυστερώ λίγο για να βάλετε και τα ακουστικά σας. Το 1993 είχαμε λοιμό στη Σομαλία το αποκορυφωμά του. Εγώ, επειδή εργαζόμουν στα ανθρωπιστικά ζητήματα, είχα την ε, δυνατότητα να εργαστώ εκεί και είδα πώ ακριβώ ε, εργάζεται και ε, ο δικό του οργανισμό, Ο Ρηθρό Για μένα ήταν η πιο πετυχημένη επιχείρηση με τη καλύτερη δυνατή λειτουργία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά. Ευχαριστώ και πάλι. Και ένα ερώτημα. Αυτός ο λοιμός τελικά αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή εθελοντών, νέων που έφερναν ε, λάδι μέσα σε βαρέλια και ε, μαγείρευαν για τις ε, υποστησμένες οικογένειες. Το ερώτημα μου είναι πώς ο Ερυθρός Σταυρός αξιοποιεί σήμερα τους εθελοντές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρολη για την παρουσίασή σας. Όπως ε, αναφέρατε, αναφερθήκατε μάλλον σε ερωτήματα προς τους πολιτικούς. Θα ήθελα και εσείς να αναφέρετε περισσότερο ότι η το αρχικό σημείο εστίαση ε, τη ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να επανεξεταστεί. Έχετε κάτι κατά νου σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βοήθεια. Είπατε ότι θα μπορούσε να δαπανηθεί με διαφορετικού τρόπου. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τα τελευταία χρόνια κατά την εμπειρία σα. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο για εμά και για την Επιτροπή μα. Αλλά αν μπορείτε να εμβαθύνετε τι ακριβώ εννοείται με αυτό, ίσω ε, και σε ό,τι αφορά άλλου μεγάλου οικονομικού φορεί, ε, για να μα βοηθήσετε και εμά στο έργο μα και στι διαβουλεύσει μα με άλλου φορεί και διεθνεί οργανισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περιμένω λίγο κι εγώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ε, Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον ίδιο και όλους τους εθελοντές που υπό δύσκολες συνθήκες επιτόπου κάνουν τόσο χρήσιμο ωφέλιμο έργο. Χαίρομαι πολύ που πέρασατε σήμερα από την Επιτροπή μας γιατί θέλουμε και εμείς να σας εκφράσουμε το σεβασμό προς ε, το έργο ε, που επιτελείται υπό τόσο δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες. Και βεβαίως σήμερα σκεφτόμαστε και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το θέμα μας, ε, βεβαίως είναι και το θέμα της ουδετερότητας. Και εγώ έχω περάσει από τέτοιες περιοχές ε, συγκρούσεων. Πώς ακριβώς ε, διατηρείται αυτή την αμερόληπτη στάση, γιατί είναι δύσκολο κανείς να τηρήσει αυτή την αρχή της ουδετερότητας. Γιατί πολύ συχνά βλέπετε και εσείς έρχεστε αντιμέτωποι με τους φορεί αυτούς τους επιθετικούς, επομένως δεν ξέρω πώς και εσείς ε, κρατάτε την αντιτερότητά σας και κάτι άλλο, που, ένα ερώτημα το οποίο μας θέσατε σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με την αναπτυξιακή βοήθεια. Εγώ είμαι υπέρμαχος ε, της ε, καλής ανθρωπιστικής συνεργασίας αναπτυξιακή συνεργασία. Όμως το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό εκεί, στις περιοχές των συγκρούσεων. Είναι δύσκολο εκεί με τα κλασικά μέσα αναπτυξιακή συνεργασία να προχωρήσει κάποιο, Δηλαδή να συνεργαστεί με τον ε, τοπικό πληθυσμό, με τους ιδιωτικού φορείς. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Όμω, το ερώτημά σας ε, μου κίνησε την περιέργεια. μήπω θα πρέπει να το επαναξετάσουμε. Και θα ήθελα να επιστρέψω το ερώτημα σε εσά Ω εμπειρογνώμονα, Μπορείτε να μας δώσετε συστάσεις και ειδικότερε συμβουλές για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μάουρε για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Αυτό το οποίο θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το θέμα των καταβλισμών προσφύγων για τους οποίους αναφερθήκατε. Υπάρχουν ήδη καταβλισμοί στη Μέση Ανατολή οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης. Επομένως δεν μπορούν να προσφέρουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στους πρόσφυγες. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο, λοιπόν, λοιπόν περισσότερο σε σχέση με την ιδέα σας να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους καταβλισμούς στη Βόρεια Αφρική. Κάβα. Ευχαριστώ. Κανείς εδώ δεν μπορεί να πει ότι δεν σέβεται ε, ιδιαίτερος ε, το έργο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Εμισελίνου. Πραγματικά θα ήθελα να πω τη σοφοροτιμή στα όσα κάνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του Σομάλιλαντ και τις ε, τελευταίες κινήσεις ε, στη Νότια Ιεμένη, έχουμε και την αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα στι Βρυξέλλε. Δύο ερωτήματα. Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ε, ο Ερυθρός Σταυρός στην Ιεμένη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι σημαίνει, τι συμβαίνει στο Σομάλιλαντ, αλλά σε ό,τι αφορά την Νότια Ιεμένη, είναι εξαιρετικά δύσκολες ε, οι συνθήκες ε, σε αυτή την ε, πλευρά της Αφρικής. Ευχαριστώ, κυρία Σουίκα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Μάουρερ για την πολύ καλή αυτή εισαγωγή. Και εγώ θα ήθελα να μέσα όσα κάνει ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Έλληνος. Το προσωπικό σας ήταν ε, παρόν ε, και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Κατά τη διάρκεια αυτού του παρεξουσμού ήταν ε, πολύ σημαντικό το έργο σας. Αναφερθήκατε σε ορισμένε περιοχές όπου υπάρχει κρίση και εκεί που παλαιότερα μάλλον είχαμε σειράξει, συγκρούσεις, πλέον πρόκειται για πόλεμο. Όμως ε, ακούσαμε και την έκκλησή σας προς εμάς, τους πολιτικούς, να συμμετάσχουμε και να βοηθήσουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να τηρήσουμε και να αρχή τα ουδετερότητας, το οποίο είναι θετικό. Όμως ένα ερώτημα που έχω είναι το εξής. δεν αναφερθήκατε σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την ε, διαχείριση των υδάτων και που δημιουργούν ε, μεγάλες δυσκολίες. Όμως υπάρχει και το ζήτημα της ε, ανεργίας θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την απασχόληση των νέων για να βοηθήσουν και παραπάνω ενώ ψάχνουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάουρερ, και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Ήθελα να σας πω ότι δούλεψα 20 χρόνια με την Ερυθράη Μισέλινο στην Λωρίδα της Γάζας και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας και τη συνεργασία μας. Ε, θέλω να κάνω δύο ερωτήματα και μία παρατήρηση. Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχει προχωρήσει το θέμα του ίδρυσης του Humanitarian Task Force που είναι νομίζω μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων την ώρα ακριβώς που πρέπει. Δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο 24ωρο που εκδηλώνεται είτε μια ανθρωπιστική κρίση είτε μια φυσική καταστροφή όπου χρειάζεται να, να εμφανίσεται ο Ερυθρός Σταυρός. Το δεύτερο αφορά το ζήτημα της ουδετερότητας. Σαφώς και όσον αφορά το ζήτημα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να τηρούμε αυστηρή ουδετερότητα και να μην αποστερούμε από κανένα την αναπτυξιακή βοήθεια. Ωστόσο, αυτή η ουδετερότητα δεν πρέπει να επεκτείνεται και στο επίπεδο του να μην προσκομίζουμε μαρτυρία για το ποιο από του δύο εμπλεκόμενου είναι ο φωνιά και ποιο είναι το θήτη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο υπάρχει μια αμφιλεγόμενη τοποθέτηση μέσα στον Ερυθρό Σταυρό ειδικά. Και το τρίτο, μια παρατήρηση δική μου είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι δουλειά του Ερυθρού Σταυρού. Είναι καλύτερα να αφήνεται σε άλλες οργανώσεις. Δηλαδή ο Ρηθρός Σταυρός έχει, α, έχει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο να παίξει. Όχι ότι η αναπτύξη είναι λιγότερο σημαντική, αλλά εν καταλαβαίνετε ότι την κρίσιμη στιγμή ο Ρηθρός Σταυρός έχει πιο μεγάλο ρόλο να παίξει. Ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot for numerous Ευχαριστώ για τα ερωτήματά σα. Ε, να πέρασω ορισμένε διευκρινήσει από πλευρά μου. Ο Ερυθρό Σταυρό έχει 14.000 ε, μέλη του προσωπικού του και όταν εργαζόμαστε στι περιοχέ συγκρούσεων συνεργαζόμαστε με την ε, τοπική κοινότητα που κινητοποιεί εθελοντέ και συνεργάζεται στενά με εμά. Ανάλογα λοιπόν με τις περιστάσει σε κάθε χώρα, έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα μεταξύ ε, εθελοντών, επαγγελματιών και τοπικής κοινότητας. Ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την εθνική αυτή κοινωνία και να επιτελέσει το έργο που δεν μπορεί να επιτελέσουν οι εθνικές αρχές. Επειδή απαιτείται διεθνής εντολή και νομιμότητα για να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένω, πάμε μετά σε πιο λεπτά ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο Ερυθρός Σταυρός. Έχουμε και τους ε, επαγγελματίες μας, αλλά γενικά σε μεγάλο βαθμό συνεργαζόμαστε με την ε, τοπική κοινωνία. Επίσης, απασχολούμε πολλούς νέους. Και εξαιτία τη αύξηση τη δραστηριότητά μα στο τελευταίο διάστημα, έχουμε κάνει και προσλήψει. Δεν ε, προτιμάμε συγκεκριμένα του ανέργου, όμω πράγματι προσλαμβάνουμε και νέου που έτσι καταφέρνουν ε, να βρουν μια δουλειά σε εμά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, αναπτυξιακή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια, όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά μέσα με διαφορετικούς ε, σκοπούς. Τώρα, το ερώτημα μου είναι αν κατά πόσο η παραδοσιακή κατηγοριοποίηση στις ε, υπανάπτυκτες, χαμηλής ανάπτυξης, μεσαίας ανάπτυξης ε, χώρες αντιστοιχεί στα όσα βλέπουμε σήμερα, όπου έχουμε θύλακες ευάλωτους θύλακε που απαιτούν ε, διαφορετική προσέγγιση. Σε κάποιες χώρες ε, είδαμε ότι έχουν διαμορφώσει νέες δομές. Είπαν ότι αντιμετωπίζουμε μία ιδιαίτερη περίπτωση. Η Ορδανία, Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Λίβανος, γειτονικέ χώρες ε, της Νιγηρίας. Δεν είναι η παραδοσιακή εξέλιξη, ανάπτυξη μάλλον ούτε η παραδοσιακή αναπτυξική βοήθεια. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια νέα δομή, ένα νέο μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να διοχετεύουμε χρηματοδότηση. Οι Ολλανδοί, για παράδειγμα, δημιούργησαν ένα τέτοιο μηχανισμό για αυτές τις ενδιάμεσες μεταβατικές καταστάσεις που είναι όλο ένα και πιο προβληματικές. Γιατί βρίσκονται στο, στις απαρχές ε, των μεταναστευτικών ροών, της αποσταθεροποίησης στις περιοχές του κόσμου και ταυτόχρονα δεν αντάσσονται στις βασικές κατηγορίες ε, ανθρωπιστική και ανεδεξιακής βοήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα, να σα πω τα εξής. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανεί να είναι ουδέτερο. Εσεί συγκεκριμένα. Είστε πολιτικοί. Δεν υποχρεούστε να είστε ουδέτεροι. Εγώ υποχρεώμαι να είμαι ουδέτερο. Η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία μας είναι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανθρωπιστική βοήθεια, για να έχουμε πρόσβαση στις πιο δύσκολες ε, συνθήκες και να ε, έχουμε και την ε, άδεια να λειτουργούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η ελπίδα μου είναι οι πολιτικοί να στηρίξουν την οδετερότητα <clears throat> του Ερυθρού Σταυρού. Εσείς, ως πολιτικοί, πολύ καλά κάνετε και λαμβάνετε θέση και θα πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε. Είναι σαφής λοιπόν η απάντησή μου. Ουδετερότητα, μεροληψία, ανεξαρτησία, εξαιρετικά κρίσιμες αξίες για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία. Εμείς καταρτίζουμε, εκπαιδεύουμε, ενσταλάσσουμε αυτές τις αξίες ε, στα 14.000 μέλη του προσωπικού μας κάθε μέρα για να γνωρίζουν όχι μόνο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, αλλά και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται τόσο ώστε και οι υπόλοιποι να τους θεωρούν αμερόληπτους και ανεξάρτητους. Αυτές είναι βασικές αξίες λοιπόν που πρέπει να τηρούν για να λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σε αυτές τις ε, πλέον δυσχερείς συνθήκες. Αν δεν είμαστε εμείς ουδέτεροι, δεν θα μπορέσουμε να παράσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ποκοχαράμ, ε, στο Ισλαμικό κράτος ή ακόμα και στο Ντονιές και το Λουγκάνσκ. Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι και να μας θεωρούν και οι υπόλοιποι ουδέτερους. Όμως εσείς ως πολιτικοί πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα έχουμε ένα τέτοιο χώρο για να μπορέσουμε να είμαστε ουδέτεροι. Όχι εσείς απαραίτητα να είστε ουδέτεροι. Αυτή είναι δική μου προτίμηση. Δεν αναφέρθηκα στις ε, κατασκηνώσεις προσφύγων στα κέντρα προσφύγων ε, στην Μεσόγειο, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός θέλει να δραστηριοποιείται όσο γίνεται πιο κοντά στην πηγή του εκτοπισμού. Γι' αυτό και κλιμακώνουμε τη δραστηριοποίησή μας ε, στην μέσα Ανατολή, στις, ε, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στην περιοχή του Τσάντ, γιατί προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο επίκεντρο της κρίσης, ούτως ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω εκτοπισμός και να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει στο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον του. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, το αναγνωρίζω δημιουργεί εντάσεις ε, μεταξύ ε, κοινωνιών ε, προέλευσης και υποδοχής. Λίβανος και Ορδανία, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. Για τις ανθρωπιστικές για τις ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα ο Ερυθρός Σταυρός τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναπτύξει ε, τις, ε, τους μηχανισμούς ταχείας ανάπτυξης που μας ε, επιτρέπει ως μηχανισμός να ξεκινήσουμε μια τέτοια λειτουργία εντός 24 ωρών με τη δυνατότητα να μεταφέρουμε 15-30 άτομα εντός 24 ωρών για να ξεκινήσει ταχύτατα μια τέτοια αντιμετώπιση μια κρίση ή μιας καταστροφή. Γι' αυτό ακριβώ ορισμένε φορέ, επειδή ακριβώ είμαστε ταχύτεροι από άλλου, είμαστε πρώτοι, φτάνουμε ε, στον τόπο μιας καταστροφής, ε, παρότι δεν ε, εντάσσεται στην εντολή μα. Για την Ιεμένη. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα όπου δυστυχώς βρούμε μόνοι μας. Ο ΙΕ δεν δραστηριοποιείται, ο ανθρωπιστικός ε, σε δεν δραστηριοποιείται στην Ιεμένη. Μόνο ε, ο Ερυθρός Σταυρός και οι γιατροί χωρίς σύνορα δραστηριοποιούνται εκεί. Επομένως, όλο το βάρος ε, πέφτει σε εμά σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίω καταλαβαίνω ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί με τις ε, μάχες και του που συνεχίζονται είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο μας. Όμως σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται σε μια επιχείρηση που είναι η πέμπτη ή η έκτη μεγαλύτερη στον κόσμο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν σημαίνει βεβαίω ότι όλοι λαμβάνουν ε, ανα πάσα στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια και αρρωγή, όμως, ακριβώς ε, χάρη στην ε, μακροχρόνια δραστηριοποίησή μας στην Ιεμένη, καταφέραμε και τώρα να βοηθήσουμε. Να σας πω τώρα κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό από αυτή την άποψη. Αρχικά, κατά τη σύλληψη της ιδέας της ανθρωπιστικής βοήθειας, είχε την έννοια της ε, προσωρινής ανακούφισης ε, των ε, επιπτώσεων μιας ε, τέτοιας κρίσης. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε αυτή την προσωρινή ανακούφιση της κρίσης και αντιμετώπιση της κρίσης. Βρισκόμαστε συνεχώς σε κατάσταση κρίσης και έτσι δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανθρωπιστικής αρρωγής και αναπτυξιακής συνεργασίας. Γιατί έχει αλλάξει ο, ο χαρακτήρας, η φύση της δουλειάς μας γίνεται όλο ένα και πιο μακροπρόθεσμος. 40 χρόνια στο Αφγανιστάν, 50 χρόνια στην Ιεμένη, δεκαετίες ε, στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό και δεν φεύγουμε γιατί κανένας άλλος ε, δεν παρεμβαίνει. Επομένω, πρέπει να εξετάσουμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα και ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς ως πολιτικοί θεωρείτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κατά πόσο οι πόροι που δαπανώνται σήμερα κατευθύνονται πραγματικά στους τομείς προτεραιότητας. Και σε επιμέρους χώρες και υπουργεία υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα, πρότυπα, νέα μέσα και νέοι μηχανισμοί για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα, μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Μάουρε, δεν είσαστε πολιτικά ουδέτερος. Μίλησατε για τον Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό κράτος. Και μίλησατε και για το Λούγκατς και το Ντόνετσκ είναι σαν να λέτε ότι οι αποσχιστικές δυνάμεις εκεί στο Λούγκατς και στον Τόνες είναι χειρότερες από τον Μπόκο Χαράμ. Κατάλαβα σωστά. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και οι προτεραιότητές μας έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι φύγονται από τις σειράξεις. Η έννοια λοιπόν της ουρετερότητος μέσα σε ένα ανθρωπιστικό πρίσμα σημαίνει ότι αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, τις ανάγκες προτεραιότητες των ανθρώπων ανεξάρτητα από το καθεστώς κάτω από το οποίο διαβιούν. Δεν συνεργαζόμαστε για να έχουμε πολιτική συνεργασία ούτε με τον Μπόκο Χαράμ, ούτε με την, το Ισλαμικό κράτος ή τις αρχές του Λουγκάνς και του Ντονέτσκ. Όχι. Ο στόχος μας είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στις τόσο δύσκολες αυτές συνθήκες. Αυτό ακριβώς είναι η ανθρωπιστική ουδετερότητα. Χρειαζόμαστε χώρο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς υπάρχει όλη αυτή η αποσταθροπή. Όλη η φιλοσοφία του Ερυθρού Σταυρού και του κινήματος του Ερυθρού Σταυρού είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα, ένας χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να δοθεί αμερόληπτη ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, χωρίς την εξάρτηση από το αν βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο μιας κυβέρνησης ή μιας ένοπλης ομάδας που έχει τον α ή τον β πολιτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο εμείς απορρίπτουμε την ιδέα του καλού ή του κακού θύματος. Τα καλά θύματα είναι αυτά που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο μιας κυβέρνησης που είναι πολιτικά ορθότερη από κάποιον άλλο. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και μόνο και αυτός είναι ο ορισμός του τι εννοούμε όταν λέμε ανθρωπιστική ουδετερότητα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και βέβαια για τις εξηγήσεις τώρα. Είναι και ο λόγος, πιστεύω, για τον οποίο ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει δραστηριότητα τόσων πολλών ετών. Όπου έχουν ανάγκη για βοήθεια οι άνθρωποι, σπέβδει χωρίς να κοιτάει προέλευση ή προσήλωση σε κάποια πλευρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που είστε εδώ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε επαφή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Kommen Λοιπόν, τώρα πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης με την ενημέρωση της αντιπροσωπείας σε σχέση με την ποσνια ερσεγοβινη Ερσεγοβίνη 21-22 Μαΐου Στρασβούργο. Γίνονται αυτές οι ενημερώσεις όπως ξέρετε διότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την αμοιβαία ενημέρωση για την αντιπροσωπεία και τις ε, εργασίες της. Ο κύριος Σπίτσου, να εδώ, παρακαλώ λάβει το λόγο. Πίκουλα. Σας ευχαριστώ, Ξιότιμοι Αξιότιμοι συνάδελφοι. 17η λοιπόν διακοινοβουλευτική συνεδρίαση δύο κοινοβούλια, 17 ευρωβουλευτές. Μαζί με τον κύριο Πρέντα, εισηγητή. Η Βοσνία είχε έξι εκπροσώπους. Επί τη ευκαιρία δεν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλους τους συναδέλφους που δεν είναι εδώ παρόντες για την συμμετοχή τους ε, στην συνεδρίαση. Είχαμε τον εκπρόσωπο της ε, υπηρεσίες για τα Δυτικά Βαλκάνια της Υπηρεσίας Εξωτερικές Δράσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπο η κυβέρνηση είχε τον επικεφαλής της Επιτροπής της Υπηρεσίας μάλλον του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και έγιναν κάποιες προτάσεις για μελλοντικές συνεδριάσεις δηλαδή συζητήσεις και απαντήσεις ε, να οργανωθούν κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι κατατέθηκαν 24 τροπολογίες σε μια κοινή δήλωση, σε ένα κοινό ψήφισμα και για το ότι η συζήτηση αυτή επέτρεψε την ομόφωνη έγκριση με βάση την αρχή, που ευκόλυνε βέβαια ιδιαίτερα, ότι οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να τροποποιήσουν κείμενα σημεία του κειμένου, ενώ οι Βόσνοι, Ευρω... οι Βόσνοι βουλευτές μπορούσαν να καταθέτουν τροπολογία. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό ψήφισμα. Και Αυτό που ακούστηκε πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια τη συνεδρίας ήταν ότι χρειάζονται αλλαγές για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Τώρα βλέπουμε ότι ε, εκφράζονται και εκκλήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων από πλευρά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και σχέση με τι γραπτέ δεσμεύσει. Επίση, ε, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με την επισήμανση ότι μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Η κατάσταση ποια είναι, η κατάσταση που θέλουμε να αλλάξει, ότι το ίμιση τουλάχιστον των πολιτών της Βοστινής Ερζεκοβίνης δεν πιστεύουν ότι μπορεί η χώρα τους να γίνει μια μέρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται βεβαίως να αντιμετωπιστούν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα παραμένουν, ζητήματα του κράτους δικαίου, ε, πρέπει να ενισχυθεί η ε, δικαιοσύνη, να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, να υπάρχει περισσότερο άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών, να καταπολεμηθεί κάθε μορφή διάκρισης και διακριτικής μεταχείρισης να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση και να γίνουν γενικά όλες οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στη Βοσνία Σεγοβίνη. Με τροποποίηση ακόμη και των πολιτικών δομών. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι από την 1η Ιουνίου του 2015 τροποποιείται το καθεστώς της αντιπροσωπείας μας, διότι τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία, για τη, συμφωνία σύνδεσης και εταιρική σχέση με τη Βοσνία, με Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν με άλλες αντιπροσωπείες, με την θέση ενισχύ της σχετικής συμφωνίας. Τα τεχνικά στοιχεία του νέου καθεστώτος αντιπροσωπείας αυτής θα διευκρινιστούν με την συνεδρίαση της διασκέψης των Πρόεδρων και αναλόγως σας ενημερώσω και εγώ. Ευχαριστώ. Σουίσα. Κυρία Σουίσα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Σουίσα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πίτσουλα. Για τις απόψεις του δεν θέλω φυσικά να επαναλάβω αυτά που είπε. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικέ οι συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών και οι εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνη έλαβαν ενεργό μέρο σε αυτέ τι συζητήσει. Θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν εκπρόσωποι της κυβέρνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνη σε αυτές τι διαπραγματεύσει, αλλά υπενθυμίζω αυτό που είπε ο κ. Σπίτσουλα. Αλλά δεν μπορούσαμε εμεί να τροποποιήσουμε τα στοιχεία τα οποία περιεχόντουσαν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε μετά από την συνάντηση. Στο τέλος λοιπόν, στην τελική δήλωση, νομίζω ότι μπορούμε να τη θεωρήσουμε ότι είναι πολύ θετική αυτή η δήλωση. Τονίζουμε τις ανάγκες για αλλαγές στην Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά επίσης τονίζουμε και τη νέα προσέγγιση που απαιτείται έναντι της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Επίσης, θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή συμφωνία σταθεροποίησης και εταιρική σχέσης με τη Βοσνία, σύνδεσης μάλλον, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις σχέσεις μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραμείνουμε στο έδαφος στο οποίο έχουμε μείνει όλο αυτό τον καιρό. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στην ανάπτυξη των σχέσεων μας με την Βοσνία Ζεγοβίνη και είναι γεγονός ότι το πρόβλημα των 50% των πολιτών που δεν θέλουν να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας οδηγήσει σε περισσότερες ενέργειες. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε η Βοσνία Ζεγοβίνη να ξαναβρει το δρόμο της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαι πεπισμένη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει η Βοσνία Ζεγοβίνη και γι' αυτό πρέπει να εργαστεί η αντιπροσωπεία μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να είστε άλλο το λόγο, γι' αυτό θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Γιατί η συμφωνία του Ντέιτον ήταν ο μόνος τρόπος να τεθεί τέρμα στον εμφύλιο πόλεμο και να οδηγήσει εφόσον υπήρχε δυνατότητα σε σύσταση ενός κράτους. Αλλά δεν είναι δυνατόν με αυτές τις δομές, αναλογικά, να γίνει ένα κράτος μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να το αντιληφθούν αυτό αναφέρεται στις συζητήσεις. Πρέπει το κράτος το ίδιο να κάνει μόνο του τα βήματα που χρειάζονται για να προχωρήσει στην ε, διαμόρφωση ενός κράτους ικανού να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά μαζί τους ώστε να το αντιληφθούν. Γιατί ένα κράτος το οποίο αδυνατεί να αναλάβει δράση, είναι ένα αδύναμο κράτος, δεν είναι δυνατόν βέβαια να επιβιώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, αλλά από τους ίδιους τους Βοσνίους. Αν και δυστυχώς, όπως είπατε, το ίμιση των κατοίκων δεν πιστεύει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δυνατότητα μάλλον ενταχθεί το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μπορούν να πιστέψουν ότι μπορεί να ε, τακτοποιηθούν τα του κράτους τους κατά τρόπο ικανοποιητικό. Όταν ε, εθνοτικές ε, αντιπροσωπείες ε, θέτουν προσκόμματα η μία στις προτάσεις της άλλης και έτσι, έτσι δεν μπορεί να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Παρακαλώ, ποιος είστε στο λόγο. Ο κύριος Πράτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποια ακόμα ερωτήματα. Ίσως ε, τα μέλη της αντιπροσωπείας μπορούν ε, να, απαντήσουν αυτά τα ερώτηματα. Πριν από λίγα χρόνια η Τουρκία ήταν πολύ ενεργή στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας πήγαινε στη Βοσνία Ζεγοβίνη κάθε δύο μήνες περίπου. Στο τωρινό τώρα χρονικό σημείο, πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε την επιρροή της Τουρκίας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Δραστηριοποιείται ακόμα η Τουρκία εκεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα των δράσεών τους και το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τη Σερβία. Ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο ασκεί η, το οποίο παίζει η Σερβία σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό αφορά και το θέμα της συνεργασίας Βοσνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν εκεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρους. Ο συγκεκριμένη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη συνέχεια των όσων είπατε για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους μετά τον Dayton, ε, έχω να επισημάνω αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές σε αυτό το σώμα, ότι η τριζωνική τρικοινοτική ομοσπονδία που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν δούλεψε. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει συνεργασία των τριών συνιστόντων ε, κρατηδίων και έχουμε αυτά τα οποία πολύ γλαφυρά περιγράψατε πριν από λίγο. Δηλαδή τον κίνδυνο να μην υπάρχει καν μια κοινή πολιτική βούληση να ενταχθεί αυτό το μόρφωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι αν αυτό δεν μπορεί να μας δώσει και κάποια παραδείγματα προς αποφυγή τη στιγμή που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε το ίδιο αποτυχημένο και καταστροφικό μοντέλο σε ένα άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατάλαβα σε ποια χώρα αναφέρεστε κύριε Θεοχάρης λέει ο, ο πρόεδρος. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ως φίλος μια σύντομη παρατήρηση. Εδώ και 20 χρόνια έχω παρακολουθήσει τα θέματα της συμφωνίας του Dayton και θυμάμαι πόση ελπίδα είχε αναποτεθεί σε αυτή την συμφωνία που στη συνέχεια δεν επαληθεύτηκε. Θυμάμαι τη Σύνοδο των Παρισίων που οδήγησε στην υπογραφή αυτού του εγγράφου και έχω φυσικά και πολύ καλή σχέση με τους ε, είπα τους εκπροσώπους των Βαλεντινίσκοφ και τον Πέτριτς που έρχονται από την Αυστρία και θυμάμαι ότι είχαμε συζητήσει στο παρελθόν για την ανάγκη επιτέλους αυτή η χώρα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Και έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια τα οποία έχουν περάσει και η εντύπωσή μου είναι, και δεν νομίζω ότι είναι μονάχα δική μου εντύπωση, νομίζω και ο κύριος Πίκουλα πιστεύω ότι θα προσυπέγραφε μια τέτοια αντιμετώπιση. Πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό συνδέεται με την δράση και του δικού μας είπα του εκπροσώπου. Είναι οι δικές του προσπάθειες που ήταν ανεπαρκείς ή στην πραγματικότητα ήταν πολύ μικρές οι δυνατότητες η χώρα αυτή να μπορέσει να προχωρήσει σε μια μεταρρύθμιση με τις δικές της δυνάμεις ή αν υπήρχαν περιορισμένες δυνατότητες να βοηθήσουμε εμείς αυτή τη χώρα να μεταρρυθμίσει τον εαυτό της με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μια δυνατότητα εν καιρό να πλησιάσει και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει Κύριε Πίκουλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω με μια φράση η οποία νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει σε όλους όσου εξέφρασαν το ενδιαφέροντό τους. Το θέμα εξακολουθεί να είναι ανοιχτό όχι μόνο για την περιφερειακή πολιτική αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική πώς μπορούμε να δράσουμε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις αλλαγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα μπορούσαμε να το συζητούμε διαμακρών και συζητώ με τον πρόεδρο Μπρόκ ότι οι αλλαγές θα πρέπει να προκύψουν ως συνέπεια εσωτερική συνένεσης και όχι ως συνέπεια εξωτερικής παρέμβασης. Οι αλλαγές θα πρέπει να προκύψουν μετά από μια εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων, μετά από εκλογές Ωστόσο, δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί εν μία νυχτή. Όσον αφορά την τουρκική επιρροή στη Βοσνία, υπήρξε η εξή σύμπτωση την ημέρα της συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Ο ε, Ερντογάν πήγε στην Βοσνία. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του για την επιρροή της ε, Τουρκίας στη Βοσνία. Δεν χρειάζεται όμως να την αντιμετωπίσουμε με φόβο τη σχέση της Τουρκίας με τη ε, Βοσνία. Εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να επεκτείνει την επιρροή της και να αλλάξει τα πρότυπά της, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξελίξεις της περιοχής. Και κατόπιν όσον αφορά τη συμφωνία, εγώ θεωρώ ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί εξαιρετικό εφαλτήριο για ε, κατάπαυση πυρός, αλλά δεν ε, μπορεί να θεωρήσουμε ότι ε, με βάση ένα τέτοιο άγγραφο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ε, οι συνέπειες της συμφωνίας ε, του Dayton πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες. Εγώ θεωρώ ότι η συμφωνία του Dayton δεν είναι προς το συμφέρον αυτών που ζουν καλά από πολιτική σκοπιά στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είπατε εκπρόσωπος Μα συγγνώμη, ο ύπατο εκπρόσωπο, ο κύριο Σίντ, ο οποίο πριν από 1,5 μήνα ήρθε εδώ στο κοινοβούλιο, ε, μίλησε μαζί μου και του είπα ότι λίγο πολύ έχει μια εξουσία αντίστοιχη με του Προέδρου Πούτιν. Έχει κάποιες εξουσίες που του επιτρέπουν να παρέμβει και να κατευθύνει τους πολιτικούς οι οποίοι πολλές φορές ερμηνεύουν λανθασμένα τα έγγραφα της ε, συμφωνίας για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε εάν αυτή η νέα στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βοσνία Ριζεγοβίνη θα αποφέρει καρπούς. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να καθορίσουμε μια καταληκτική προθεσμία. Φέτος πρέπει να δούμε αν θα υπάρξουν ε, ε, μέχρι το τέλος του 2015 κάποιες ε, ε, ελπίδες βάσει της νέας προσέγγισης. Ευχαριστώ. Μετά από τις προετοιμασίες που έχουν γίνει, ίσως ο κύριος Πρέντα τώρα μπορεί να μας αναφέρει τη δική του άποψη ο Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά ήμουνα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ε, είχαμε τους κοιόδης εισηγητές. Εγώ θεωρώ ότι η συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος, η 17η ε, συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βοσνίας Ερζεγοβίνης, όπου ανέχτηκαν την παρουσία μου επειδή ήμουν εισηγητής, δεν είμαι μέλος της συγκεκριμένη αντιπροσωπείας. Ήταν όμως μια πολύ καλή ε, συνάντηση. Τα μέλη του Κοινοβουλίου της Βασνίας Ερζεγοβίνης ήταν από διάφορες πολιτικές οικογένειες, επομένως είχαμε πλήρη κάλυψη και θεωρώ ότι ήταν και μια ευκαιρία να περιγράψουμε ε, με τους πιο απλούς όρους τις θέσεις μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η θέση των βουλευτών από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ήταν ότι τους ενδιαφέρουν και οι ευρωπαϊκές υποθέσεις, ε, έγιναν και ε, αρκετές συζητήσεις για το τι σημαίνει το τάδε ή το δίνα και πρόκειται για συνεδριάσεις οι οποίες ε, ήταν αρκετά ουσιαστικές. δεν είχαμε αυτό που βλέπουμε και σε άλλες ε, συνεδριάσεις αντίστοιχες, ε, κάποιες επικρίσεις ίσως ε, στις παρεμβάσεις. Πιο πολύ σταθήκαμε σε εξηγήσει και νομίζω ότι το τελικό συμπέρασμα είναι στην ίδια άγουσα της έκθεσης που εγκρίναμε και εμείς εδώ τον Απρίλιο και νομίζω ότι κατοπτρίζει πολύ καλά τις θέσεις ε, των δύο πλευρών από τον Οκτώβριο και μετά. Μετά από αυτή τη νέα σύνθεση των συναντήσεων ε, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες ανταλλαγές απόψεων που θα έχουν και κάποιες επικριτικές ε, ε, πτυχές και θα είναι έτσι και πιο ζωηρές ε, λόγω αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Πίτσουλα για τις προσπάθειες που έκανε ώστε να ε, υπάρξει μια καλή συνάντηση στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ και ο Πρόεδρος. Έχουμε 15 λεπτά για διάλειμμα. η πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας θα έρθει σε περίπου 15 λεπτά, λέει ο πρόεδρος Μπροκ.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

Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση μα λοιπόν. Έχουμε το θέμα 6 στην ημερήσια διάταξη. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω την πρόεδρο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατρίν Πάντσα. Τη συνοδεύει ο Υπουργό των Οικονομικών, ο Υπουργό των Εξωτερικών και η Υπουργό της Εθνικής Οικονομίας. Και η υπουργό των Κοινωνικών Υποθέσεων επίση. Καλώ ήρθατε λοιπόν σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνομιλήσουμε μαζί σας σήμερα. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εξελίξεις στη χώρα σας. Και με μεγάλη χαρά παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικές με την ολοκλήρωση των προσπαθειών για την Εθνική Συμφιλίωση στον Πανγκουί. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Το ταχύτερο δυνατό. Ιδιαίτερος χαίρομαι για το ότι υπέγραψαν οι ένοπλες ομάδες με την κυβέρνηση, τη συμφωνία για, την, για τον αφοπλεσμό, την ε, επιστροφή των ενόπλων στον πολιτικό βίο και τη συμφιλίωση. Ελπίζουμε ότι έτσι μπορεί να τελειώσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας και ελπίζουμε ότι η κυβέρνησή σας αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις, οι ένοπλες ομάδες θα μπορέσουν να ακολουθούσουν το δρόμο μιας ειρηνικής μετάβασης. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στις ε, δυνάμεις της μετάβασης. Κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε για την υλοποίηση του σχεδίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαιτέρως παρακολουθεί τις εξελίξεις στην κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Θα γνωρίζετε ίσως ότι συνάδελφοι της Υποεπιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας υπό την κυρία Φωτσίκα ε, επισκέφθησαν τη χώρα σας. Είναι εδώ παρόντες ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα της ασφάλειας μαζί σας. Ο κύριος Κούλογλου επίσης είναι εδώ, εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, που επίσης παρακολουθεί τα θέματα αυτά και θα θέλαμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για τις εξελίξεις στη χώρα σας. Έτσι ώστε να είμαστε και εμείς σε θέση να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας προς τη χώρα σας και την προσήλωσή μας στον αγώνα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχετε το λόγο. Euh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Κυρίε και κύριοι, εξέχουσες προσωπικότητες, είναι μια μεγάλη τιμή για μένα και έχει ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα για μένα η ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ σε εσά εκπροσώπους του σημαντικού αυτού του υψηλού θεσμικού οργάνου που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας ευχαριστήσω για όλες τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβετε <clears throat> υπέρ της διαδικασίας ειρήνευσης, εξασφάλισης της ασφάλειας, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οικονομικής ανάκαμψης της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Η συνεχή σας δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή το πνεύμα αλληλεγγύης που έχετε επιδείξει, το οποίο διατρέχει όλες τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είναι ακριβώς το έμβλημα της Ευρώπης, που είναι ένας από τους κύριους φορείς ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και υπέρμαχου των οικουμενικών αξιών και αρχών. Κυρίες και κύριοι, με τον να σήμερα την Επιτροπή σας, την τόσο σημαντική και έγκυρη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θέλω εκ μέρους της χώρας μου να συναντήσω την Ευρώπη και τους λαούς που εσείς εκπροσωπείτε. Η Ευρώπη είναι ένας ιστορικός εταίρος για μας. Εδώ και πολλές δεκαετίες παρακολουθείτε τα εκτενομένα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε όλους τους τομείς. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών η χώρα μας η κεντροαφρικανική δημοκρατία <clears throat> έχει διατρέξει μια σειρά από σοβαρές κρίσεις, τις πιο σοβαρές ίσως σε όλη την ιστορία της. Γενικευμένη ανασφάλεια, χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση, κατάρρευση του οικονομικού ιστού, παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων, καταρακωμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλα αυτά οδήγησαν στην απόγνωση για όλους τους πολίτες της χώρας μου. Κυρίες και κύριοι, από τη στιγμή που ανέλαβα τα ενία της μεταβατικής κυβέρνησης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου ως μητέρα του έθνους μου να ακούσω τις εκκλήσεις, τις απέλπιδες εκκλήσεις του λαού μας και να προσπαθήσω να κινητοποιήσω τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσει το λαό μας. Έχουν γίνει πολλές εκκλήσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη και προς όλους τους διμερείς εταίρους μας, καθώς και τους πολυμερείς διεθνείς φορείς. Έχουμε καταφέρει να θέσουμε στο επίκεντρο των παγκόσμιων ανησυχιών και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο έχω έρθει και προσωπικά στις Βρυξέλλες τον προηγούμενο έτος για να ζητήσω τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας ώστε να ευδοκιμήσει η διαδικασία ειρήνευσης και η διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για το γεγονός ότι βρήκαν ευήκοα ότα αυτές οι εκκλήσεις. Υπήρξε μια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καταλάβει το μέγεθος των διακυβευμένων και έχει ξεκινήσει μια σειρά από με το ε, να δημιουργήσει και ένα ταμείο σταθεροποίησης το Ταμείο Μπεκού, το οποίο έχει σαν στόχο την σταθεροποίηση της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ε, επαναφοράς των εθνικών και περιφερειακών αρχών της ε, εξασφάλισης των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών στη χώρα με Όπως σας είπα, η κεντροαφρικανική δημοκρατία πηγαίνει καλή, πολύ καλύτερα. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα μου παρά το γεγονό ότι παραμένει ακόμα ιδιαίτερα ευάλωτη η κατάσταση. Σιγά σιγά επανέρχεται η ειρήνη στον Μπαγκή και σε ορισμένα τμήματα της χώρας μου. Σε ανθρωπιστικό επίπεδο, ο αριθμός των ατόμων που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι έχει μειωθεί. Από ένα εκατομμύριο που ήταν εκτοπισμένοι πριν από ένα έτος, έχουμε, έχουμε κατέβει στις 450.000 μονάχα. Είναι ένας ποσοτικός δείκτης πολύ σημαντικός. Σε οικονομικό επίπεδο, <clears throat> από μείον 35% από ύφεση 35% στην κορυφή της κρίσης πριν από ένα έτος, έχουμε περάσει σε οικονομική ανάπτυξη 1,6% για το 2014 και προχωρούμε προς το 4 ή 5% το 2015. Επιπλέον, η αύξηση των οικονομικών μας πόρων έχει γνωρίσει μια ανάπτυξη κατά 100%, μια αύξηση κατά 100%. Ήταν τεράστια λοιπόν και πάρα πολύ σημαντική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαν να καρποφορήσουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Γι' αυτό και πάλι θέλω να τονίσω και πάλι την ευγνωμοσύνη του λαού της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για όλες τις προσπάθειες που κάνατε για να μπορέσετε να βοηθήσετε τη χώρα μου να βγει από την κρίση. Σε επίπεδο ασφάλειας ήσασταν παρόντες. Η κινητοποίηση πάνω από 500 εκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσει να υπάρξει ε, βοήθεια στο ματηρικό μου λαό, ο οποίος αντιμετώπιζε πολλαπλές πηγές βίας, ήταν πολύτιμη. Ο λαός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας εκτιμά ιδιαίτερα το ρόλο που διαδραμάτισε η ΦΟΣ στην διαδικασία αυτή. Θέλω λοιπόν Formal. Θέλω να τονίσω το ρόλο των Ευρωπαίων στρατιωτών που έπαιξαν νευραλγικό ρόλο στη διαδικασία εξασφάλισης της ασφάλειας στην πόλη του Μπαγκή από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Θέλω να κύψω την κεφαλή μου ενώπιον των νεκρών της ΕΟΦΟΡ. Ήταν ένα παράδειγμα πάρα πολύ σημαντικό για το λαό μας, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα στη χώρα μου η οποία προσπαθεί κάθε μέρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Πολίτες που στρατιώτες που ήρθαν από χώρες που ήταν εμπόλεμες πριν από μερικές δεκαετίες τώρα αγωνίζονται υπέρ της ειρήνης. Η Ευρώπη είναι δίπλα μας με την ε, ε, υποστήριξη της μεταρρύθμισης της δυνάμεις ασφαλείας της χώρας μου. Σε οικονομικό επίπεδο επίση ήσασταν αρρωγή. Με την υποστήριξη προς τον προϋπολογισμό όμως που ήταν απαραίτητη για να μπορέσει να ανακάμψει και να σταθεί στα πόδια της η οικονομία μας που είχε καταρρεύσει. Σε πολιτικό επίπεδο επίση ήσασταν παρόντες μέσω της συμμετοχής σας στην Διεθνή Ομάδα Επαφής που μας βοηθήσατε ώστε τα παιδιά μας να μπορέσουν να βρουν μια λύση σε αυτή την κρίση και να σταματήσει αυτή η αναμόχλευση και η συνέχιση του εσωτερικού μίσους. Δεν μας εγκαταλείψατε ποτέ. Με τη μόνιμη παρουσία σας μας δώσατε μια παρηγορία, μας δώσατε και πάλι το χαμόγελο, μας επιτρέψατε να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά μας. Βοηθήσατε και περιθάλψατε τους ασθενείς μας. Δώσατε υποστήριξη και σχολικό υλικό στα παιδιά στους μαθητές. Δώσατε βοήθεια στους ε, καταβλισμούς των προσφύγων και των εκτοπισμένων για να μπορέσουν όλοι αυτοί να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά τους. Σε εσά, εκπροσώπους της Ευρώπης που βρίσκεται εδώ, θέλω λοιπόν από το βάθος της καρδιάς μου να εκφράσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ε, ευγνωμοσύνη μου και την αναγνώριση όλου του λαού της κεντρικής της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας για τη βοήθειά σας. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά είναι πάρα πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Η κεντροαφρικανική δημοκρατία βασίζεται σε όλους σας για να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε στην ε, εκταμείευση των κονδυλίων για να ξεκινήσουν τα απαραίτητα σχέδια στη χώρα μας. Είμαστε δεσμευμένοι στο να δημιουργήσουμε καινοτόμους μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν την απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας. Αυτή η αποτελεσματικότητα και αυτή η διαφάνεια είναι μια θεμελιώδης απέτηση του λαού μας που δεν θα δεχτεί πια τις διαδικασίες και τις ενέργειες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κράτους στο παρελθόν. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα πρέπει να ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία της για το όφελος των παιδιών μας. Θα πρέπει να ιδρύσουμε ένα νέο κράτος, να έχουμε μια νέα, ένα νέο συμβόλαιο με τους πολίτες μας, να ξεπεράσουμε τα ερήπια του παρελθόντος, να εξασφαλίσουμε τη συμφιλίωση όλων των πολιτών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, ώστε να ξαναβρούμε την κοινωνική συνοχή και την συλλογική ζωή που ήταν στο παρελθόν το κέντρο της δύναμής μας και της υπερηφάνειάς μας κυρίε και κύριοι. Από τότε που είμαι επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης έχω θέσει την ασφάλεια, την ειρήνη, την εθνική συμφιλίωση και την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στο κέντρο των προτεραιοτήτων μου. Χωρίς όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική επανίδρυση του κράτους. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις βασικές επιδιώξεις του λαού μας, ο οποίος χρειάζεται δικαιοσύνη αλλά ζητά και μια νέα μορφή δημοκρατικής διακυβέρνησης που να βασίζεται στην ευθύνη, στην ακαιρεότητα αυτών οι οποίοι είναι στην εξουσία. Προς την κατεύθυνση αυτή, μετά την υπογραφή των, της συμφωνής, συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στην Πραζαβίλ, οργανώσαμε και ήταν επιτυχές αυτό, ε, δημοψηφίσματα ουσιαστικά σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις κοινότητες της χώρας μου. Και με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε να συλλέξουμε και να αντιμετωπίσουμε τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες του πληθυσμού μας. Έχουμε δημιουργήσει το Εθνικό Φόρουμ του Μπαγκή από τις 4 έως 11 Μαΐου που μας έδωσε δυνατότητα να οργανώσουμε μια διαβούλευση και ένα ζωντανό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των ζωντανών δυνάμεων του λαού μας μεταξύ αυτών των δυνάμεων του στρατού και της κυβέρνησης μετάβασης. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δεν θα οδηγήσουν σε απογοήτευση, γιατί έχουμε καταδείξει με το φόρμα αυτό ότι οι χθεσινοί εχθροί στην κεντροαφρικανική δημοκρατία μπορούν να χαράξουν μαζί το δρόμο του αύριο και από κοινού να ανοίξουν το δρόμο της ελπίδος την ελπίδα να ζήσουμε από κοινού ειρηνικά, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, να προωθήσουμε το κράτος δικαίου, το σεβασμό της δικαιοσύνης, την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών, τον αγώνα κατά της ατιμορρησίας, το δικαίωμα για την προσωπική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη, το σεβασμό για τη ζωή, την ελπίδα για όλους τους πολίτες της Κεντρικοαφρικανικής Δημοκρατίας να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους την ε, μοίρα τους και να μπορέσουν να εκλέγουν ελεύθερα τους ηγέτες τους και οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το έθνος. Από αυτή την έννοια πάντοτε έχω ανάγκη από την ε, πολυδιάστατη βοήθεια της Ευρώπης για να μπορέσω να αρθώ στο ύψος αυτών των προκλήσεων. Εκλογές, παραδείγματι, όπου χρειάζεται μια επιπλέον ε, προσπάθεια. 18 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κενό Στο δημοσιονομικό κενό επίσης, στο δημοσιονομικό έλλειμμα, όπου χρειάζεται ακόμη να βρεθούν 21 εκατομμύρια δολάρια. Στην ασφάλεια επίσης, η πρόκληση σε σχέση με, την, με τον αφοπλισμό, την αποκινητοποίηση, την, ε, τον επαναπατρισμό. Χρειαζόμαστε 67 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια δολάρια. 67 εκατομμύρια. Κυρίε και κύριοι, απευθύνω έκλειση σε όλα τα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να βοηθήσουν το λαό μου να σταθεί στα πόδια του και να μπει στο δρόμο της συμφιλίωσης, της ε, ανάπτυξης κοινωνικής και οικονομικής. Είμαι βέβαια ότι θα σταθεί και πάλι στα πόδια της κεντροαφρικανικής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και θα αγωνιστώ με όλους μου τις δυνάμεις, ώστε μετά τη μετάβαση να υπάρξουν νέα θεμέλια, να αναθεμελιωθεί μια νέα κεντροαφρικανική δημοκρατία, ορθή, υπερήφανη, αποφασισμένη, ευημερούσα, μια κεντροαφρικανική δημοκρατία της οποίας ο κάθε γιος και κάθε θυγατέρα θα είναι σε σχέση συμφιλίωσης μεταξύ τους και θα μπορούν να ορίσουν μόνοι το μέλλον τους και τις ανάγκες τους. Ζήτω η συμφιλία, ζήτω η φιλία μεταξύ Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και Ευρώπης. Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλική σας ε, ακρόαση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εγώ για τα σοφά σας λόγια. Μας δίνουν μεγάλη ελπίδα. Έχω μια ερώτηση και εγώ πριν αρχίσει η συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν σχεδιασμοί και σχέδια για τις περαιτέρω κινήσεις σε σχέση με το εκλογικό ημερολόγιο για τις προεδρικές και τις κουλευτικές εκλογές. Απάντηση. Η εκλογική διαδικασία ε, προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα βάση του μεταβατικού προγράμματος που φτάνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2015. Εν ώψη αυτή τη ε, ημερομηνία, χρειάστηκε να ομολογήσουμε ότι θα μπορούσαν από ηλική άποψη και μόνο να διοργανωθούν αυτέ οι εκλογέ. Επομένω, προβλέψαμε ένα νέο ε, διάστημα έξι μηνών με εκλογέ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και μετάβαση τη εξουσία ε, στι νέε αρχέ τον Αύγουστο και προβλέψαμε και συγκεκριμένο προπολογισμό. Σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους ε, για να γίνουν αυτές οι εκλογές μέσα στην προθεσμία και επομένω το Φόρουμ του Μπαγκή αποφάσισε η, διεθνή κοινότητα αλλά και η εθνική κοινότητα που έχει αναλάβει την ε, ε, ενέργεια των εκλογών να συγκεντρωθούν και να αποφασίσουν μία νέα ημερομηνία. Δεν μπορούμε όμως να ξεπεράσουμε το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Δεν είχε προβλεφθεί ούτε για την χώρα μου, ούτε για τους υπόλοιπους εταίρους μας να ε, αναβάλουμε επάπειρον ε, την μεταβατική αυτή κυβέρνηση. Να την διατηρήσουμε μάλλον. Η περιφερειακή η οργάνωση ε, έχει αναλάβει να επικυρώσει το χρονοδιάγραμμα και είπαμε ότι θα γίνουν εκλογές το αργότερο το Δεκέμβριο του 2015. Όταν επανέλθουμε λοιπόν στον Παγκή, θα μοιράσουμε ακριβώς αυτή την περίοδο με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να γίνουν οι εκλογές. Αυτά έχω να σας πω για το θέμα των εκλογών κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκούλογλου εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας, τα πολύ θερμά σας λόγια και ενθαρρυντικά. Ε, ε, Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία ειδικού ενδιαφέροντο για εμά στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ανθρωπιστικές ανάγκες, το Ευρωπαϊκό Καταπίστευμα Μπεκού και η μελλοντική αναπτυξιακή συνεργασία με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. με τον 10 ο Αναπτυξιακό Ταμείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι πάνω από το ίμιση του πληθυσμού της χώρας αυτή θεωρείται ότι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 600 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια θα πρέπει να κινητοποιηθούν βάσει του σχεδίου στρατηγικής ανταπόκρισης όμως μέχρι τώρα μόλις 11% αυτού του ποσού έχει διοχετευθεί προς τη χώρα. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω το εξή. Είστε αισιόδοξοι ότι οι βασικές ανάγκες του λαού σας ε, θα πληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας έχει φύγει τώρα από το επίκεντρο της προσοχής ε, των ε, μέσων ενημέρωσης και αυτό έχει και τον κίνδυνο για μια φορά ακόμη να ξεχαστεί η χώρα σας. Δεύτερο σημείο, σε ό,τι αφορά το καταπίστευμα Μπεκού. Ή το, το Μπεκού σημαίνει ελπίδα. Η ελπίδα ήταν λοιπόν και νέοι επιπρόσθετοι εταίροι να ε, συμμετάσχουν στο καταπίστευμα, να αυξήσουν τους πόρους και να διευκολύνουν τη συνεργασία. Επομένω, εσείς, ε, κυρία Πρόεδρε, τι άποψη έχετε για αυτό το καταπίστευμα και αν θεωρείτε ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και των προσδοκιών σας, αν υπάρχουν άλλοι δωρητές που θέλουν, ε, χορηγοί που θέλουν να συμμετάσχουν και Τρίτο, η Επιτροπή μας κλείνει τον προγραμματισμό του 11ου Ευρωπαϊκού Νοτοξιακού Ταμείου. Το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Αφρικανική Δημοκρατία θα έρθει για έγκριση από την Επιτροπή στο δεύτερο εξάμεινο φέτος και έτσι οι συζητήσεις με τη κυβέρνησή σας ελπίζω να προχωρήσουν θετικά. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιους τομείς θα θέλατε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί. Το Κοινοβούλιο μας θεωρεί ότι ιδίω η παιδεία είναι μοχλός ανάπτυξης και ότι η βασική υγειονομική περίθαλψη πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, αναπτυξιακή μας συνεργασία. Βάσει τελευταίων στοιχείων η εθνισμότητα των παιδιών κάτω από 5 ετών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι 129 προς χίλιους, που είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Μόλις 10% των γυναικών έχουν ε, κάποιο είδους ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το ποσοστό αναλφαβητισμού είναι πάνω από 56% στο γενικό πληθυσμό. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς το μεταβατικό συμβούλιο, η προσωρινή κυβέρνηση δηλαδή, εμπλέκεται και συμμετέχει στις ε, συζητήσεις για αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ, κυρία Φωτίγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ε, εκ μάλλον της Υποεπιτρεπής ε, ασφάλεια και Άμυνας θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ε, που υποδεχθήκατε την αντιπροσωπεία μας στην Κεντροφρυγανική Δημοκρατία. Επισκεφθήκαμε τη χώρα σας το Φεβρουάριο του 2015 και πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θετική και συγκινητική αυτή η αποστολή η επίσκεψή μας στη χώρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά, αλλά να ευχαριστήσω και τους ε, εκπροσώπους όλων των ε, επιπέδων διακυβέρνησης της χώρας σας. Υπήρχαν και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν, γιατί εκπροσωπήθηκαν και όλες οι θρησκευτικέ πεπιθήσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ επικοδομητική ε, στάση τους ε, στην, ε, στην αντιπροσωπεία μας. Χαιρόμαστε που η γενική αντίληψη σε ό,τι αφορά την επιτυχία της αποστολής μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ήταν τόσο θετική. Ο ρόλος αυτής της αποστολής συναδέλφωσης, γεφύρωσης και μετάβασης στην ε, αποστολή Μινούσκα. Ήταν εξαιρετικά σημαντική. Και μάλιστα κατάφερα ε, να συναντήσω και τους συμπατριώτες μου Πολωνούς ε, στρατιώτες που και αυτοί συμβάλλουν στην σταθεροποίηση της περιοχής. Κυρία Πρόεδρε, χαιρόμαστε που μετά από αυτή την αποστολή είχατε αυτό το πολύ σημαντικό επίτευγμα του Φόρουμ Μπαγκή, που μάλιστα υπέγραψε την ε, συμφωνία DDRR. Ε, υπεγράφει από την ε, πλειονότητα των στρατιωτικών ε, ομάδων, και συγκεκριμένα της ΕΛΕΚΑ και την Αντιβαλάκα. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη κατά τη γνώμη μας. Θα μπορούσατε κι εσείς να αναφερθείτε περαιτέρω στην ανάγκη ανάληψης νέων ενεργειών, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοδοτικές ανάγκες για την επιτυχή και κατάλληλη διενέργεια εκλογών στην καταπληκτική Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ του ΕΛΚ σας καλωσορίζω εδώ και θα ήθελα καταρχάς ε, να σας συγχαρώ για τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίσατε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα σας. Σας εύχομαι καλό κουράγιο για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία έρχεται να συμπληρώσει αυτή που σας έθεσε ήδη ο πρόεδρός μας και ε, στην οποία έχετε ήδη απαντήσει για τις εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους. Εγώ θα ήθελα από αυτά που ήδη διευκρινίσατε να ξέρω Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή για τις εκλογές. Θεωρείτε ότι θα πρέπει καταρχάς να διοργανωθούν προεδρικές εκλογές και μετά κοινοβουλευτικές ή ε, Ξέρετε ότι αυτό είναι θέμα το οποίο συζητάμε πάντα όταν υπάρχει πολιτική κρίση και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας ε, για το πώς ε, θα πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές. Ε, δεύτερον, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τη συμφωνία η οποία προέκυψε προσφάτως στον Μπαγκουή για, από το διάλογο αυτό από το Υπουργείο Άμυνας και των διαφόρων ένοπλων ομάδων, Εξ όσων γνωρίζω, ένα από τα στοιχεία τα οποία αποφασίστηκαν ήταν να ε, ενταχθεί κάποιος από αυτές τις ένοπλες ομάδες ε, στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχει ε, πρόβλεψη και για κατάλληλο προπολογισμό για αυτή τη διαδικασία και αν έχετε αριθμιστικά στοιχεία. Πόσοι άνθρωποι από αυτές τις ενοπλές ομάδες θα ενταχθούν σε ενοπλές δυνάμεις. Υπάρχουν ε, κάποιες προβλέψεις, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για αυτή την ευαίσθητη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας και για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ ε, την ε, Πρόεδρο για την παρουσία της. Ε, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι οι στόχοι αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης, της οποίας προεδρεύει, είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εσωτερική διαδικασία ειρήνης εντός της χώρας και να ε, έχει ως στόχο την ανάπτυξη. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα και είναι και πολύ άριθμα προβλήματα τα οποία κρεμούν και ίσως με τη δράση σας καταφέρετε να μετριάσετε απλώ τα αποτελέσματα και όχι να ε, επιλύσετε την πρόβλημα, το πρόβλημα μεταξύ των διαφόρων φυλών που μάχονται μεταξύ τους. Θα ήθελα να ξέρω και την άποψή σας επί του ζητήματος. Υπάρχει ένας καταβλισμός προσφύγων στη χώρα που είναι από τους μεγαλύτερους καταβλισμούς στο Μπατάγκαφό και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς μας μιλήσατε και μας είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα συμφωνία. Εγώ φρονώ ότι αυτή η νέα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σίγουρα θα πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρώ ότι πρέπει και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε να συμφωνήσετε ότι χρειάζεται και πιο στεναρή δράση από πλευράς μεταβατικής κυβέρνησης ιδίως ε, όχι απλώς ε, για τη διεξαγωγή των εκλογών, αλλά για να ξεκινήσει και αυτή η ειρηνευτική διαδικασία και να επελυθούν κάποια προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά στη χώρα σας. Ε, επισητιστική ασφάλεια, ασφάλεια εν γέννη, προστασία των εθών πολιτών και διάσωση όλων αυτών που πεινούν. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας για το πώς μπορείτε να υπερβείτε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν στήσει το λόγο ακόμα 7 συνάδελφοι. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μα. Έτσι λοιπόν, εάν μπορέσει ο καθένα σα να περιοριστεί στο ένα λεπτό παρέμβαση, θα αφήσουμε λίγα μόνο λεπτά, γύρω στα 5-6 λεπτά στην ε, κυρία Πρόεδρε για να απαντήσει. Σα παρακαλώ πολύ πολύ θερμά, ένα λεπτό μόνο καθένας, ο κύριο Μισελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και μια και έχω μόνο ένα λεπτό, θα το αξιοποιήσω όσο περισσότερο μπορώ. Μια και έλαβα μέρος ως ειδικό απεσταλμένος της ε, γαλλοφωνής στην ε, συνέλεση αυτή, θέλω να ενημερώσω ότι το φόρουμ του Μπαγκή ήταν τεράστια επιτυχία, χάρη στη, στα χαρίσματα και την προσήλωση της κυρίας Πρόεδρου. Πρέπει να το πούμε αυτό Χρειάζεται να την υποστηρίξουμε και θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδώσει αυτή την έκκληση ώστε να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις από τους χορηγούς. Ο κίνδυνος και η πρόκληση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι ακριβώς αυτό. Να μπορέσει να συλλέξει επαρκή οικονομικά μέσα, στο το εξαιρετικό αυτό σχέδιο που έχει ετοιμάσει, που έχει κυρία ε, σαν Παπάντζα να υλοποιηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που θα βρούμε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε το ειδικό δικαστήριο που είναι στοιχείο της καταπολέμησης της ατιμορρησίας, πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια για την αποκατάσταση και την ε, ε, επιδιόρθωση όλων αυτών των υποδομών του κράτους που είναι η δικαιοσύνη, η αδέκαστη, η εκπαίδευση, τα σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Πρέπει λοιπόν και απευθύνω έκκληση προς τη δική μας πλευρά να ε, παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση διαρκώς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν καλύτερη κινητοποίηση πόρων. Πρόεδρος, μα ξεπεράσετε και το χρόνο σας όμως. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω σου ειδικά, Κύριε Σεβαλός. Ήμουν μεταξύ εκείνων που ήθελαν να επικεντρωθούν περισσότερο στην ε, κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Ε, με την επίσκεψη μπορέσαμε να παρατηρήσουμε τα γεγονότα μαζί με την κυρία Φουτσίγκα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με την EU4, και της συνέχισης της παρουσίας δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το άλλο είναι αυτό το πρόβλημα των διάτριτων συνόρων στα ανατολικά της χώρας και του λαθρεμπορίου όπλων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι λύση έχετε προβλέψει για τα θέματα αυτά. Και επίσης σε σχέση με την κατάσταση εδώ στη Δύση. Γιατί ξέρετε πολλέ φορέ εδώ στη Δύση βλέπουμε μια εικόνα διαθρησκευτικών συγκρούσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται μερικέ φορέ η κατάσταση, ενώ εγώ δεν είχα την ίδια αντίληψη από την επίσκεψή μου. Μπορείτε λοιπόν να μα επιβεβαιώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω στο ερώτημα αυτό το οποίο μόλις αναφέρθηκε. Πράγματι, υπήρξαν αυτές οι διαθρησκευτικές οι διαδογματικές ε, συγκρούσεις. Ποια ήταν, ποιος ήταν ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών και η προσπάθεια που κατέβαλαν για την συμφιλίωση επίσης σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας. Είπατε ότι θα ενσωματωθούν οι πολιτοφυλακές στον Εθνικό Στρατό. Βλέπετε εδώ να είναι χρήσιμο το να υπάρξουν κάποιες ε, συμβουλές από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, του, ή από την ε, Αφρικανική Ένωση, από χώρες που έχουν περισσότερη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Κύριο Σπαρνιό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω εδώ μαζί με την κυρία Φώτιγκα, την κυρία Σεμπάγιο, τον κύριο Ντανζόν ήμουνα στην αποστολή της Υποεπιτροπής Ασφάλειας που ήρθε στον Παγκή στις 21 Φεβρουαρίου πρέπει να πω και δεν θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι αλλά πρέπει να σας πω είχαμε μια πολύ θετική εντύπωση όχι μόνο από εσά και την προσωπικότητά σας από τον τρόπο με τον οποίο έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία συμφιλίωσης και ανοικοδόμησης της χώρας σας που ήταν τελείως κατεστραμμένη. Δύο ερωτήματα ο στρατός. Αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ανοικοδόμησης <clears throat> που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και τη σταθερότητα. Όταν όμως ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών ε, ομάδων μέσα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με ποιο τρόπο θα δημιουργηθεί αυτός ο νέος στρατός, με ποια στάδια θα γίνει αυτό. Επίσης, <clears throat> η διεθνής κοινότητα έχει τονίσει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ατιμορρησία για κάποιους ηγέτες της Αφρικής που ακόμα και έξω από την δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής θα πρέπει να έρθουν ενώπιον της δημοκρατίας. Τι ρόλο θα παίξει αυτό στη διαδικασία συμφιλίωσης γιατί δεν είναι ένα ανώδυνο πρόβλημα μονάχα. Κύριος Τένοκ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ εξ ονόματος ομάδος ECR να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι είσαστε και η πρώτη γυναίκα που έχετε αυτό το υψηλό αξίωμα ως επικεφαλής κράτους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στη μεταβατική αυτή διαδικασία. Για το θέμα της δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης της ατιμορρησίας. Είσαστε, ε, έχετε την ε, πεποίθηση ότι θα μπορέσει να γίνει η διαδικασία αυτή σε εθνικό επίπεδο. Η Amnesty International ανέφερε το ένα πρώην πρόεδρο και ένα ηγέτη μιας ομάδος ως ε, πιθανούς κατηγορούμενους. Πιστεύετε ότι μπορούν να απαγγελθούν καταγορίε εναντίον αυτών ή πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να υπάρξει ε, προεδική χάρις προς αυτούς ώστε να μπορέσουν και οι αντάρτες να ενσωματωθούν ομαλά σε αυτή τη νέα δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Επίσης ξέρετε ότι το Ισλαμικό κράτος είναι ενεργό σε πολλά μέρη της Αφρικής, έχετε πρόβλημα με τον τζιχαδισμό και το Ισλαμικό κράτος προσπαθεί να προσελκύσει και να στρατολογήσει μαχητές για τη Συρία και το Ιράκ και επίση αναφερθήκατε στο ρόλο τη υποπεριφερειακή οργάνωση ΕΚΑΣ τη Δυτική Αφρική. Μερικοί από αυτού του φορεί έχουν αναπτύξει και τα δικά του δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι μπορούν να σα βοηθήσουν και εσά και την Αφρικανική Ένωση στο να φέρετε ενώπιον τη δικαιοσύνη του ε, υπεύθυνου για εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, κύριε Κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως θα θέσω το ερώτημά μου. Και θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε ένας προλαλής σας. Για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές τις συγκρούσεις. Ο επίσκοπος του Μπαγκή είπε ότι πρόκειται για μια πολιτικο-στρατιωτική ε, σύγκρουση. Δεν είναι μονάχα θέμα εξουσίας, αλλά ήταν και θέμα χρημάτων, πλούτου. Μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε Ποιε είναι οι συγκεκριμένες αιτίε αυτή τη πολιτική και οικονομική σύγκρουσης και αν υπάρχουν κάποιες χώρες της δύση οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτή τη σύγκρουση. Υπήρξαν και από τις δύο τώρα από παρατάξεις παρα, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων από στα θέματα τη Αφρικανική Ένωση. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό και πώ προχωρούν οι ανακρίσει για αυτό το θέμα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια τη μελλοντική διαδικασία συμφιλίωσης. Μπασίρ, τελευταίο ανοχίστατο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρα για την παρουσία, Πρόεδρο, για την κυρία σας... παρουσία σας εδώ. Και θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, αν ήταν ζήτημα ισχύω και οικονομικό και όχι θρησκευτικό, τότε γιατί τόσο σημαντικό αριθμό μουσουλμάνων μπήκε επίση σε, σε αυτού του καταβλισμού ε, και έχασε τη ζωή του. Επίση, ε, τι μέτρα έχουν ληφθεί για να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι στι ε, περιοχέ τους και σε ό,τι αφορά τα ε, μουσουλμανικά τεμένη και την οικοδόμησή τους, ε, τι συμβαίνει εκεί. Γιατί θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι ένα καλό μοσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. από τον αριθμό των ε, βουλευτών που πήραν το λόγο, βλέπω πραγματικά και διαπιστώνω το μεγάλο ενδιαφέρον σας ε, για τη χώρα μου. Οι παρατηρήσει ήταν πολύ διαφορετικέ μεταξύ του. Αφορούσαν και την ανθρωπιστική κατάσταση, την πολιτική κατάσταση και την ε, ε καταπολέμηση τη ατιμορρησία. Θα ήθελα να ομοδοποιήσω τι ε, απαντήσει μου για να μην απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. σε ό,τι αφορά την κατά παρέμβαση ε, που αναφέρεται στο καταπίστευμα Μπεκού, ε, έχει λάβει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τον ανθρωπιστικό τομέα, με όλη την ε, διαδικασία αρρωγής και ανακούφισης των προβλημάτων του πληθυσμού. Όλα αυτά αποτελούν τη βασική μας μέρημνα στο καταπίστευμα Μπεκού τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί αφορούν κυρίως την παιδεία, την υγεία, την ε, γυναική επιχειρηματικότητα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, νομίζω ότι ο πρώτος ε, ομιλητή είπε ότι πάνω από το ίμιση του πληθυσμού ε, χρήζει ανθρωπιστικής βοήθειας, που ήταν τεράστιο ο αριθμό και θα πρέπει και εμεί κάτι να κάνουμε για να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό έχω έρθει κι εγώ εδώ, εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένε ανάγκε, υπάρχουν σημαντικέ προσδοκίε από την πλευρά του λαού μου και εγώ δεν έχω τα μέσα να αντιμετωπίσω αυτές τις, για να καλύψω αυτές τις ανάγκες, γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση στην διεθνή κοινότητα. πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη που πάντα μας βοήθησε και να πούμε Ορίστε, έχουμε πόρους που έχουμε διοχετεύσει στο Μπεκού. Εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας τώρα μαζί και με την ε, συνδρομή άλλων χωρών ευρωπαϊκών ή μη, γιατί έχουμε και ε, συνεισφέροντες που δεν είναι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βρισκόμαστε λοιπόν εδώ και ελπίζουμε η παρέμβαση της Ευρώπης να μην περιοριστεί μόνο στις ε, δηλώσεις προθέσεων, αλλά σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ε, εκταμείευση αυτών των πόρων, για την πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι και ο σκοπός της έκκλησης που απευθύνουμε. Το ποσοστό θνησιμότητας που αναφέρει, και τα ξέρουμε όλα αυτά τα δραματικά στοιχεία, την δραματική κατάσταση την οποία βιώνει ο πληθυσμός μας. Επειδή ακριβώς θέλουμε να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση, πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο να ζητήσουμε τη βοήθεια των υπολείπων για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ε, ε, κατάσταση, το βιωτικό επίπεδο, αλλά και μορφωτικό και, και τα λοιπά του πληθυσμού μας. Σε ό,τι αφορά ε, τις μεταβατικές αρχές, βεβαίως ε, και έχουν αφοσιωθεί σε αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο όραμα της κυρίας ε, Σαμπά Παντζά, είναι ένας ε, μοχλός μόνο ε, αυτό το πρόσωπο για την πρόοδο της χώρας μου. Έχω ένα όραμα για τη χώρα μου, αλλά εκεί θέλω να συμμετάσχουν όλες ε, οι θετικές ε, δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα μου και έτσι φτάσαμε στην λαϊκή διαβούλευση όπου ο κόσμος πραγματικά εξέφρασε ε, τις επιθυμίες και προσδοκίες του και έτσι φτάσαμε στο φόρουμ του Μπαγκή. Καταφέραμε να αφήσουμε κατά μέρος το παρελθόν και να κοιτάξουμε μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να βελτιωθούν τα πράγματα. Βεβαίω δεν πρόκειται να επιληθούν ω διαμαγεία όλα τα προβλήματα. Εκεί θα είναι τα προβλήματα. Όμω από κοινού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ή ε, να τα μετριάσουμε τουλάχιστον. Όταν είπα ότι και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πάει καλύτερα, είναι επειδή ακριβώς ξεκινήσαμε από ύφεση 37%. Μπορείτε να φανταστείτε. Για μένα το 1,5% τώρα είναι εξαιρετικό. Είναι ένα μεγάλο βήμα που έχουμε ήδη κάνει. Είμαστε στο 1,6 και οδεύουμε προς τα 4. Αν είμαστε και αισιόδοξοι μπορεί και παραπάνω. Πάνε καλά τα πράγματα λοιπόν. Προσπαθούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα για να ξεφύγουμε αυτήν την κατάσταση. Όμως δεν πρόκειται βεβαίως τα προβλήματα αυτά μεταξύ των ε, τοπικών ε, κοινοτήτων, ε, τα οικονομικά, τα κοινωνικά ζητήματα να επιληθούν. Απλώς πραγματικά θέλουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα, τα επόμενα βήματα. Από σήμερα το πρωί μόνο για αυτό μιλώ, για τα επόμενα βήματα. Ήδη πριν από ένα χρόνο όταν είχα έρθει, είχα ε, παρουσιάσει τις προτεραιότητες. Δημοσιονομική βοήθεια, στήριξη της εκλογικής διαδικασίας, ε, της ε, ανακούφισης των προβλημάτων του πληθυσμού, μαζί με τον ε, ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς είχαμε εντοπίσει ακριβώς ε, αυτές τις ανθρωπιστικές ε, ανάγκες. Ένα χρόνο μετά δεν έχουμε λάβει ακόμα, δεν έχουν ταμιευθεί αυτά τα ποσά. Υπάρχουν δηλώσεις προθέσεων, αλλά πολύ λίγες ενέργειες. Επομένω, επανέρχομαι στους εταίρους μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, υπήρξαν δεσμεύσεις, δήλωση προθέσεων. Τώρα θέλουμε πράξεις. Αυτό είναι και το νόημα της παρουσίας μου εδώ. Τώρα για τις εκλογές. Να σας πω ότι η εκλογική διαδικασία αποφασίστηκε κοινή συνενέση από τις επιμέρους δυνάμεις και θα γίνουν από κοινού όλες οι εκλογές, προεδρικέ και βουλευτικές. Όμως πριν από τι εκλογές θα έχουμε και το συνταγματικό δημοψήφισμα, γιατί εκτιμήσαμε ότι μετά από όσα τα όσα πέρασε η χώρα μας θα πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα και να ε, εντάξουμε σε αυτό στοιχεία που να επιτρέπουν ε, την συμβίωση, την ελληνική συμβίωση, αλλά και τον κοσμικό χαρακτήρα, τον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δυσκολίες που είχαμε στις επιμέρους περιοχές και να ε, επανεβεβαιώσουμε την βούλησή μας να πάμε στην αποκέντρωση, ούτως ώστε οι ε, τοπικές αρχές να είναι πιο αυτόνομες ε, και να εκμεταλλεύονται ακόμα και τους πόρους μας προς όφελος του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική συμφωνία, ανέφερε ότι ήταν ένα πρώτο βήμα προς τις ε, προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν από κοινού. Είναι μια κοινή λοιπόν απόφαση των ενεργών δυνάμεων του έθνους πολλά ερωτήματα αφορούσαν τις ένοπλες δυνάμεις ε, και ένοπλες ε, τέτοιες ομάδες. Σε ό,τι αφορά τις ένοπλες ομάδες και την ε, διείσδυσή τους στις ένοπλες δυνάμεις, στις στρατιωτικές ομάδες ο στρατός, η αστυνομία, οι δασονόμοι, οι πυροσβέστες, όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να απορροφήσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Τι είπαμε λοιπόν, να πάρουμε χιλιάδες ε, ε, στρατιώτες ε, των Αντιμπαλάκα ή των Σενεκά να τους βάλουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Όχι θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα τον καθένα για να δούμε τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται σε κάθε σώμα για να ενδυναμώσουμε και πάλι τις ε, δυνάμεις μας, τα σώματά μας, για να γίνουν πραγματικά επαγγελματικά σώματα που ανταποκρίνονται στις, στα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά την άμυνα και την προστασία. Αυτό είναι ένα βήμα στο οποίο θα προχωρήσουμε. Ήδη το έχουν εξετάσει αυτό οι ενεργέ δυνάμεις στην συμφωνία που υπεγράφει με τις ένοπλες δυνάμεις, ομάδες μάλλον, ότι δέχονται να αφήσουν ε, τα όπλα και να απορροφηθούν από τις ε, ένοπλες δυνάμεις. Πριν τις εντάξουμε όμως θα πρέπει να έχουμε ένα όραμα για τον στρατό μας. Τι στρατό θέλουμε, ποια είναι η μορφή που θέλουμε να του δώσουμε λέμε θέλουμε 5.000 ε, άτομα για παράδειγμα. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να δούμε τους απόστρατους, τους ε, τραυματίες πολέμου, τους λιποτάκτες. Πρέπει να καθαρίσουμε αυτό τον στρατό από αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτό και όταν θα έχουμε μια κοινή θεώρηση του στρατού που θέλουμε, μετά θα μπορέσουμε να περάσουμε στην ε, απορρόφηση αυτών των πρώην μαχητών. Αυτά συζητήσαμε και στο φόρουμ του Μπαγκή, αλλά και σε άλλους ε, πιο συγκεκριμένους ε, φορείς. Αυτό είναι, αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δούμε πιο ξεκάθαρα τι θέλουμε σε ό,τι αφορά την ε, άμυνα και προστασία. Γι' αυτό προηγουμένως απίθυνα έκκληση όχι μόνο για την περίοδο που αναφέρθηκε, αλλά και για μετά αυτή την περίοδο ότι θα χρειαζόμαστε την συμβουλευτική στρατητική αποστολή UMAM για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων μετά. Ευχαριστώ τον ε, Πρωθυπουργό Λουί Μισελ για την έκκλησή του. Θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση. Αρκετά μιλήσαμε αρκετές δηλώσεις προθέσεων κάναμε, τώρα πραγματικά πρέπει να δράσουμε. Να υπάρξει ενεργό στήριξη τη κεντροαφρικανική δημοκρατία. Χωρί αυτή την ενεργό στήριξη δεν μπορούμε να περάσουμε στι εκλογέ και αν δεν έχουμε εκλογέ θα βρισκόμαστε και πάλι σε αυτή την μεταβατική περίοδο που δεν είναι θετική για την χώρα μου. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η μετάβαση. Η μετάβαση είναι πάντα προσωρινή. Πρέπει τώρα να περάσουμε σε νέε δομές και θεσμούς. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Άλλα ερωτήματα αφορούσαν ε, τον θρησκευτικό ή μη χαρακτήρα της σύγκρουσης. Αρχικά η σύγκρουση δεν ήταν θρησκευτική, ήταν διακοινωτική πολιτική. Όμως είχε και θρησκευτικές προεκτάσεις, το αναγνωρίζουμε. Η ίδια, στην απαρχή λοιπόν δεν βρισκόταν το θρησκευτικό στοιχείο, μετά όμως ε, πολλοί αξιοποίησαν ε, τη θρησκεία για να επιτύχουν τους στόχους τους. Και βεβαίως ε, βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο πλέγμα θρησκευτικών και κοινοτικών ομάδων, κοινοτήτων μάλλον, αλλά η βασική αρχή και αιτία δεν είναι θρησκευτική. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για θεμελιώδη θρησκευτικά ζητήματα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την ατιμορρησία ε, και την δίωξη των ε, παλαιών ε, τέος προέδρων, νομίζω ότι έχουν ληφθεί μέτρα εναντίον συγκεκριμένων προσώπων μέχρι την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, το κλείσιμο κάποιων λογαριασμών πρέπει να ε, σεβαστούμε τις δεσμεύσεις που λαμβάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Δεν γίνεται και να αποφασίζουμε το ένα και μετά να κάνουμε το άλλο. Αποφασίστηκε ότι πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον ορισμένων προσώπων για τα όσα έχουν κάνει. Πρέπει και εμείς να το σεβαστούμε λοιπόν. Και οι Κεντροαφρικανοί είχαν πει ότι στη, κατά τη διάρκεια του διάλογου η ατιμορρησία δεν θα υπάρξει θέλουμε να περάσουμε τη συμφιλίωση χωρίς νόμους να γίνει αυτό μέσω της δημορρησίας. Πάντα υπήρχε αμνηστία κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας, αλλά στο τέλος ε, πάντα είχαμε τα ίδια, μια αρνητική σπήρα. Και η αμνηστία τελικά δεν έφερε αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να συνεχίσουμε και να αφήνουμε να πληρώνουν τα θύματα της ενέργειας εκείνων οι οποίοι στον ε, αιώνα των άπαντα θα επωφελούνται από την ατιμορρησία και θα επαναλαμβάνουν τις πράξεις τους. Με την λαϊκή λοιπόν αυτή, με τα λαϊκά αυτά δημοψηφίσματα, τη λαϊκή διαβούλευση, ήταν εξαφές το μήνυμα ότι ήταν πρόημο το να επιτρέψουμε να επανέλθουν ορισμένοι προκειμένου να έχουμε ανοιχτή στάση και, και δεκτική προς όλους. Έπρεπε αυτοί να μείνουν απ' έξω προς το παρόν. Και για ορισμένους υπήρξε ζήτημα για το φόρουμ του Μπαγκή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το κάνουμε στο δυνατόν πιο ανοιχτό προς τους πάντες. Νομίζω ότι εξάτλησα τις ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί. Εκτοπισθέντες, πρόσφυγες. Για τους εκτοπισθέντες υπάρχει το ανθρωπιστικό πάνω απ' όλα η ε, κατεπίκουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν το ανθρωπιστικό ζήτημα, το ζήτημα της υγειονομικής ε, περίθαλψης κτλ. Ε, πρέπει τώρα, αφού ξεπεράσαμε το στάδιο αυτό, να κοιτάξουμε την πραγματική ανόρθωση, την ανοικοδόμηση, τη δυνατότητα να επανέλθουν στις περιοχές όπου ζουν παλιά οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι το όραμά μας τώρα. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να φύγουν από τα στρατόπεδα, από τους καταβλισμούς των εκτοπιστέντων, όπου ζουν ήδη, και να τους στηρίξουμε να επανέλθουν στις περιοχές ε, καταγωγής τους. Βεβαίω αυτό χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε κάποια βασικά στοιχεία. Μερικές φορές ε, δεν χρειάζονται και πολλά, ξέρετε. Ένα-δύο κομμάτια καραβόπανο και δύο πάσαλοι για να στήσουμε μία σκηνή ή να φτιάξουμε μια είσοδο σπιτιού. Είδατε ποια ήταν η κατάσταση στο μπάνκι όσοι ήρθατε στο αεροδρόμιο όπου πολλές φορές λινάτσες, απλά ούτε καν λινάτσες, ε, σάκι είναι το μέσον με το οποίο στεγάζονται οι άνθρωποι αυτοί ε, μέσα στη λάσπη σε συνθήκες ε, φρικτές σε σχέση με την ε, υγιεινή. Θέλουμε να ξεφύγουν από αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να, για να τους κάνουμε να ξεφύγουν από αυτό να τους ξαναπετάξουμε πίσω συνθήκες της άγριας φύσης. Πρέπει να τους προσφέρουμε επαρκείς συνθήκες. Αυτό σημαίνει χρήματα βεβαίως. Και είμαστε πεπισμένοι ότι και οι εταίροι θα συνεχίσουν να μας ε, βοηθούν. Έχω πιστεύω εξαντλήσει τις ερωτήσεις, κάποιες είχαν κοινά θέματα. Ευχαριστώ για την έκδηλη, για το έκδηλο ενδιαφέρον σας, για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει και ο Πρόεδρος Μπροκ. <clears throat> Οι, τα χειροκροτήματα δείχνουν την μεγάλη εμπιστοσύνη που τρέφουμε προς το πρόσωπό σας σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας ειρήνευσης και δημοκρατικής εξέλιξης στη χώρα σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και έχετε την απόλυτη υποστήριξή μας. Ευχαριστώ πολύ για την έλευσή σας. Έχουμε τώρα το υπόλοιπο, την κρόαση για την Κίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως με την ακρόαση για την Κίνα, γιατί έχουμε μόνο 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Γιατί μετά έχουμε την ψηφοφορία πρέπει να ξεκινήσει εν καιρός. Εν καιρός, λέγω. This Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω με την ακρόαση για την Κίνα. Θα ήθελα να σας πω όμως επίσης, πριν από τρεις εβδομάδες έλαβε χώρα η 400η επέτειος. Τεσσαρακοστή λέγω επέτειος της ε, σύναψης επισημών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ήταν με, το, με την ευκαιρία αυτή η κυρία Μογκερίνη στο Πεκίνο και έλαβε μέρος σε ένα υψηλό επίπεδο στρατηγικό διάλογο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Κίνα βρίσκεται σε μια νέα φάση βλέπουμε ποιες είναι οι νέες επιλογές της σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν μονάχα ένα παράδειγμα αυτό η Τράπεζα Ασιατικών Επενδύσεων, η AIIB, η συμμετοχή στην Τράπεζα BRICS της Κίνας επίσης, η συμμετοχή της σε θέματα παγκόσμιας διακυβέρνησης που θέλει να ασκήσει κάποιο ρόλο. Επομένως αυτά είναι θέματα τα οποία εμπλέκουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρου διότι ο κόσμος αλλάζει. Και το μέγεθος της Κίνας σε οικονομικό επίπεδο θα έχει και αντίκτυπο σε πολιτικό επίπεδο. Επομένως, εμείς θέλουμε η Κίνα να αναλαβεί περισσότερες ευθύνες για την επίλυση των κρίσεων στον κόσμο μας. Και όχι μονάχα προς το δικό της όφελος, αλλά προς το γενικό συμφέρον θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ελπίζω λοιπόν ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα υπό την ε, ε, ηγεσία του Γιώ Λάινεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει όλες αυτές τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Κίνα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Λάινεν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να είμαι σε αυτή την ακρόαση. Βέβαια 45 λεπτά δεν μπορούν να αρκέσουν για να τόσο τεράστιο θέμα, για να είμαι σύντομος, η στρατηγική ε, εταιρική σχέση με την Κίνα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η ουσία, ποια είναι τα σχέδια που εμπλέκονται. Αυτό είναι λοιπόν το κομβικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Μετά από 40 χρόνια διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο του εμπορίου και μόνο θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια πιο συνολική εταιρική σχέση που να περιλαμβάνει όχι μόνο τον οικονομικό στίβο αλλά και τα πολιτικά θέματα. Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για τη διμερή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, αλλά επίση και για τι παγκόσμιες ευθύνε που επομίζεται η Κίνα, όπω αναφέρατε, η παγκόσμια σταθερότητα, η συνεργασία για την προάσπιση των κοινών αγαθών σε πλανητικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην ε, Ανατολή, στην Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Ευρώπη Όλα αυτά είναι πολλές ευκαιρίες να συνεργαστεί η Ευρώπη με την Κίνα για τα θέματα ειρήνης και σταθερότητας. Και φυσικά έχουμε και το θέμα της ανάπτυξης και της συνδετικότητας, μια κοινή αφρικανική στρατηγική για τα θέματα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε το Σεπτέμβριο, η υπεράσπιση κοινών αγαθών όπως είναι η ενεργειακή πόρη και η αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής και φυσικά πώς θα αντιμετωπίσουμε το νέο κόσμο του διαδικτύου, την ε, προστασία δεδομένων και την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Είναι μια, σειρά, μια πλειάδα θεμάτων λοιπόν που θα εμπλέξουν και εμάς και την Κίνα στο μέλλον. Για να είμαι σύντομο λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι αμοιβέ, απειλέ, αλλά μπορούν να διαδραματίσουν ένα συμπληρωματικό ρόλο και γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερα να συζητήσουμε αυτήν την στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και προσβλέπω σε αυτά που θα μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας οι οποίοι θα προσθέσουν και στοιχεία για την έκθεση που συγγράφει ο κύριος Μπέλτερ για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Φρανκ και έχει το λόγο καταρχήν. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους δύο πρόεδρους που μου δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ για περίπου 10 λεπτά για τη σύγχρονη Κίνα. Τι θα κάνω σε αυτά τα 10 λεπτά θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι η Κίνα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε με απλούς χαρακτηρισμούς, όπως για παράδειγμα ότι είναι απλώς μια κομμουνιστική χώρα που ε, έχει ξεφύγει λίγο, ε, αλλά η Κίνα έχει διάφορες ε, ε, πτυχές, τις οποίες ε, σε κάποιες περιπτώσεις αναγνωρίζουμε και σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων απόψεών της, ώστε να καταλάβουμε και την πολιτική, αλλά και την προσέγγιση που ακολουθεί η κινέζικη κοινωνία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα της Κίνας είναι το γεγονός ότι η Κίνα είναι μια χώρα σαν την πρώην Σοβιετική αιώνια ένωση, ε, ένα σοσιαλιστικό κράτος ε, το οποίο ε, κυβερνάται από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό μια περιγραφή σημαντικών πτυχών της πολιτικής και της κοινωνίας της Κίνας. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ακόμα τα ενία. Εγώ θα μπορούσα δεν να σας πω ότι είναι περισσότεροι οι ε, ισχύς του τώρα από ό,τι πριν από 20 χρόνια και έχει κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει τη μορφή της Κίνας και να ενισχύσει και την διοίκηση και να δημιουργήσει μια διοίκηση που θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη διακυβέρνηση της κινέζικης κοινωνίας. Αυτή είναι και η πρώτη μου παρατήρηση, ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις αν θέλετε, σε ένα σοσιαλιστικό κράτος και σύστημα, στην πραγματικότητα ενισχύουν το ένα το άλλο, δεν είναι αντιφατικά στοιχεία, ούτε έρχεται το ένα σε αντίθεση με το άλλο. Η ιδέα ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις οδηγήσουν σε δημοκρατική μετάβαση ε, σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε λανθασμένα τα στοιχεία. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πλήρως τα ενία ε, σε... Ε, αντίθεση με όλες τις άλλες δομές που υπάρχουν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η Κίνα είναι μια πλήρως αποκεντρωμένη κοινωνία και έχει ένα πλήρως αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα. Ε, σε κάποιο βαθμό ε, μοιάζει και αντίστοιχο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές από τις επαρχίες της Κίνας ε, και ε, μέσα σε αυτές οι νομαρχίες και οι δήμοι ε, σε μεγάλο βαθμό είναι αυτόνομες μονάδες ε, που έχουν ίδια οργάνωση και οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι υπεύθυνοι για όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης, ε, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημαρίας του λαού και ε, μία σειρά από πολιτικών που είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μεγάλο βαθμό ελάχιστη κεντρική άμεση σχέση έχει η κεντρική διοίκηση ε, στο Πεκίνο. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει στη σύγχρονη Κίνα και είναι και μια αρχή διακυβέρνησης και μια αρχή της ε, κυβέρνησης που επανεπιβεβαιώνεται συνεχώς από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι δηλαδή ένα πολυτερχικό σύστημα στο οποίο το κεντρικό, ε, η κεντρική κυβέρνηση αποφασίζει τα πάντα και όλοι κάνουν αυτό το οποίο τους έχουν διατάξει. Οι Κινέζοι βέβαια πέρα από ε, κομμουνιστική χώρα είναι και μία ε, οικονομία ελεύθερης αγοράς τύπου Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, όλοι γνωρίζουμε τι μεταρρυθμίσεις έγιναν, τι έχουν φέρει, την οικονομική ανάπτυξη που δημιουργήθηκε, η οποία είναι ε, χωρίς προηγούμενο παγκοσμίω. Δεν χρειάζεται να σας δώσω εγώ τα στοιχεία, τα βλέπουμε από διάφορες πηγές, αλλά είναι σαφές ότι οδήγησε σε ένα τομέα της κοινωνίας, ο οποίος αναπτύσσεται συνεχώς, και ε, είναι καπιταλιστικός εκφύσεως, τον κυβερνούν οι αγορές. Αλλά δεν είναι ε, εντελώς ανεξάρτητο από το κράτος. Κάποιες πτυχές ίσως είναι ανεξάρτητες, αλλά κάποιες άλλες είναι απόλυτα συνδεδεμένες με το κράτος ε, σε όλες τις μορφές της διοίκησης και εντός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και αυτό το οποίο γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα κρατικές επιχειρήσεις, περίπου 100 επιχειρήσεις, οι οποίες ε, έχουν καθοριστεί από την κεντρική κυβέρνηση ως η λύθη της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, αντίθετα από ότι ε, θα συνε... μάλλον όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Η Κίνα όμως δεν είναι μόνο ο συνδυασμός μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας και μια καπιταλιστικής αγοράς. Η Κίνα ε, είναι όλο ένα και περισσότερο, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό και ίσως πρέπει να το αναφέρουμε, ε, κάτι ε, αντίστοιχο των αφροκανικών ε, ε, απολυταρχικών καθεστώτων, αυτές τις κοινωνίες που έχουμε κυρίως σε τοπικό επίπεδο, και δεν περιορίζονται όμως μόνο σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα ε, μαζί με τη διακυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αρχίζει να είναι και, ολοένα και πιο έκδηλο. Υπάρχουν διάφορες εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες επιβάλλουν πολιτικές, υπάρχουν τοπικοί ε, αρχηγοί των οργανώσεων και ε, υπάρχει φυσικά και συνδικαλιστικό έγκλημα στην κορυφή. Προσφάτως ο κύριος Λιώχαν εκτελέστηκε για διαφθορά και εκβιασμό, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στο Πεκίνο. Σίγουρα η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεωρούν ότι απειλεί το Κομμουνιστικό κράτο και το Κομμουνιστικό Κόμμα παρά το γεγονό ότι το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετέχει. Μια τέταρτη εικόνα της Κίνας ένα τέταρτο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να το αναγνωρίσουμε εμείς. Είναι κάτι το οποίο ομοιάζει πολύ σε μια κοινωνία, με μια πολύ ισχυρή κοινωνία των πολιτών, με ένα πολυφωνικό πολιτικό σύστημα, ένα πολιτικό κλάδο αν θέλετε, ε, στον οποίο δεν υπάρχουν μόνο πρώην δημοκρατικές οργανώσεις και μηχανισμοί που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, αλλά επίσης και η ίδια κοινωνία των πολιτών μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και τοπικές ε, οργανώσεις. Το τελευταίο πρόσωπο, και με αυτό θα σταματήσω, είναι μια Κίνα που αρχίζει να μοιάζει ε, με μια χώρα σαν τη Σιγκαπούρη. Ένα καλοπροέλερετο πολιταρχικό σύστημα το οποίο βασίζεται σε κοινωνική χειραγώγηση περισσότερο της κοινωνίας και όχι τόσο σε ε, διακυβέρνηση της κοινωνίας. Είναι μια κοινωνική διακυβέρνηση, διαχείριση αν θέλετε. Ε, θα σταματήσω τώρα, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για τον ε, νέο επικεφαλή, τον Ξησυγκίνγκ, αλλά ίσως θα αφήσω χρόνο για ερωτήσεις. Ο καθηγητής Μαν, η καθηγήτρια μάλλον κυρία Μεν, η οποία θα μιλήσει για τη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνες. Το θέμα μου είναι η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνας και εγώ δεν θα αντιμετωπίσω μονάχα τις δύο αυτές πλευρές. Θα το δούμε και, και τις διμερείς σχέσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα και την Ανατολική Σχέση, μένω στο Βέλγιο εδώ και 20 χρόνια και πριν ε, είχα. Διέμενα μάλλον στην Κίνα, επομένω έχω δει τα πράγματα και από τι δύο πλευρέ. Αν δούμε τα πράγματα από πλευρά ιδεολογία, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικού συστήματο, προβλημάτων ε, και τα λοιπά, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η σχέση. Αλλά αν το εξετάσουμε από την σκοπιά των συμφερόντων, ε, βλέπουμε ότι η Κίνα τώρα γίνεται πιο πλούσια, έχει περισσότερη ισχύ, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να συνεργαστούμε μαζί της και να τη βοηθήσουμε και την ίδια στη διαδικασία ένταξής της στο διεθνές ε, σύστημα. Και εκεί υπάρχει ευρύ ε, πεδίο συνεργασία. Όπω είπε και ο κύριο Πίκε, λοιπόν, υπάρχουν πολλέ πτυχέ και στι ε, σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Επομένω, όταν εξετάζουμε τι ε, σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, πρέπει να πούμε ότι και από την πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη σκοπιά τη Κίνα υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει, διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικοί στόχοι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια πάντα θέλει και προτίθεται να μεταμορφώσει την Κίνα, να την αλλάξει. Από το πρώτο έγγραφο πολιτικής που είχε εκδοθεί το 1995 μέχρι και σήμερα έχει την ιδέα να αλλάξει την Κίνα. Αν δείτε στον ιστό τοπό ε, της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κίνα λέει ότι υποστηρίζουμε την μετάβαση της Κίνας σε μια ανοιχτή κοινωνία βάσει του κράτους του δικαίου και ε, τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή είναι η αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσεχές μέλλον. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει 100 χρόνια. Από την άλλη πλευρά ε, η Κίνα λέει ότι θέλει ισότιμη μεταχείριση. Επίση ώρε λοιπόν να γίνονται συζητήσεις. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν οι δύο πλευρές έχουν διαφορετικά μηνύματα ε, στο διάλογο που γίνεται μεταξύ τους. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, γίνεται λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση η Κίνα στι σχέσεις τη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλε χώρε, αλλά και με την διεθνή κοινότητα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να αλλάξει κανεί ε, την Κίνα, να εκπληρώσει ε, του επιμέρου στόχου του. Και έτσι θεωρώ ότι είτε μα αρέσει η Κίνα είτε όχι, βρισκόμαστε σε ένα κόσμο συνύπαρξης είτε μισούμε την Κίνα είτε όχι, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την Κίνα. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε με την Κίνα και να αυξήσουμε ε, την κοινή μας ωφέλεια. Επανέρχομαι τώρα στην στρατηγική ε, εταιρική σχέση με την Κίνα. Είναι στρατηγική εταίρη και ναι και όχι μπορεί να απαντήσει κανείς. Ναι γιατί είναι και σημαντική στην ε, παγκόσμια διακυβέρνηση, πρέπει να συνεργαστούν σε πολλά στρατηγική σημασία ζητήματα. Από την άλλη όχι γιατί είναι πολύ διαφορετική δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αλληλοκατανόηση μαζί τους μέχρι τώρα. Πιο πρόσφατα όμως ένας Αμερικανός καθηγητής προετοίμασε, εκπώνησε μία ε, έκθεση για αυτό το θέμα και ε, έθεσε τον τίτλο «Επικοδημητικός ρεαλισμός. Σχέσεις με την Κίνα». Αν εγώ έπρεπε να ορίσω τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, θα πρότεινα τον τίτλο «Επικοδοματικός φιλελευθερισμός για κοινά συμφέροντα». Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποστολή να αλλάξει την Κίνα, ε, στόχος είναι η διεύρυνση του διαλόγου, θεσμικών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για να την ε, παροτρύνουμε να κινηθεί πιο κοντά προς την οικονομία της αγοράς. Όμως αυτό θα γίνεται βαθμιδών και με αμοιβή εμπιστοσύνη και με κοινά συμφέροντα. Αλλιώ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, είναι αναντικατάστατη σε αυτόν τον κόσμο και από εμπορική σκοπιά. Ο εμπορικό όγκο είναι 1 δι ευρώ ανά ημέρα και η Κίνα είναι η δεύτερη σε μέγεθος ε, γεωργική αγορά για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και με βάση του προγράμματο υποδομών Juncker οι κινεζικέ επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Ευρώπη και σε ό,τι φορά την ε, διμερή συμφωνία επενδύσεων ε, έχουν ολοκληρωθεί πέντε γύροι διαπραγματεύσεων, τον Ιούνιο θα έχουμε τον έκτο και η Κίνα είναι διατεθειμένη να απορροφήσει ή μάλλον να ε, υιοθετήσει περισσότερους διεθνεί κανόνες και να προωθεί σε αυτή τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ γνωρίζετε ότι σε ό,τι αφορά και την ε, αϊφόρα ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή κτλ. πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα να συνεργαστούν, να βρεθεί μια λύση για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα όμως και πάλι να τονίσω ότι για το σκοπό της συνεργασίας με την Κίνα ένας ε, βράχη και πρόθεσμο στόχο θα πρέπει να είναι και μέσο πρόθεσμο θα είναι η συνεργασία και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εργαστούμε για να αλλάξει ε, η Κίνα και να γίνει μια κοινωνία βάση του κράτου δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω βράχη και μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, συνεργασία. Τέλο, για την ε, προώθηση τη εταιρική σχέση, Θα έχω ορισμένες προτάσεις εδώ. Πρώτον, πρέπει θα υπάρχει οικοδόμηση θεσμών, διάλογος ε, και συνεργασία. Μετά, ε, κατάρτιση περισσότερων εμπειρογνωμόνων στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Και τρίτον, επαφές σε επίπεδο βάσης, δηλαδή ε, ανταλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο αν θέλετε και ενίσχυση του πολιτισμικού διαλόγου. Και τέλο, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον, αλλά όχι στο Πεκίνο. σω έχει έρθει η ώρα και το Κοινοβούλιο να εξετάσει ε, να ε, διαμορφώσει μια τέτοια μόνιμη αντιπροσωπεία στο Πεκίνο. Ευχαριστώ, κύριο Βόουτερ. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα κάνω μια πολύ συνοπτική ε, παρουσίασε από τη βάση του σχεδίου μελέτης μας που είχαμε κάνει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιέχει μερικές κέρυες συστάσεις και προτάσεις. Καταρχήν, η εξωτερική πολιτική της Κίνας πρέπει να αντιμετωπιστεί με, βλέποντας την αλληλεξάρτηση και το άνοιγμα της Κίνας προς τον έξω κόσμο. Παρά την ε, εικόνα που δίνει προς τα έξω, το στόχος της Κίνας ακόμα, το τι θέλει να κάνει με όλο αυτό το άνοιγμα παραμένει ανοιχτό. Από τη μια μεριά η πολιτική της ε, Κίνας φαίνεται να εξαρτάται από την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές προκλήσεις. Αλλά συγχρόνως αυτή η πολιτική οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από μια περιστασιακή και πραγματιστική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό της αβεβαιότητας, η εξωτερική πολιτική της Κίνας έχει παρουσιαστεί ως πιο αποφασιστική τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στην ε, ρητορική της Κίνας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και στις δράσεις της. Τέσσερα σημεία σχετικά. Πρώτα απ' όλα, η Κίνα έχει καταδείξει τη θέλησή της να ασκήσει στρατιωτική δύναμη πέραν στρατιωτική ισχύ, πέραν και των συνόρων της, όταν διάσωσε Κινέζους εργαζόμενους στα μέσα της κρίσης της Λιβύης, αλλά επίσης και με την συμμετοχή της στην ενέργεια κατά της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής. Δεύτερον, η Κίνα όλο και περισσότερο δείχνει να έχει ένα αποφασιστικό ρόλο στο να διεκδικεί κυριαρχικότητα στο ανατολικό και νότιο κινέζικο πέλαγος και έχει χρησιμοποιήσει και εθνικιστικές κορώνες για να υποστηρίξει την ε, διεκδίκησή της. Τρίτον, η Κίνα έχει ξεκινήσει να διαμφισβητεί μερικούς από τους κύριους φορούς διακυ... διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ζητώντας εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ή δημιουργώντας εναλλακτικούς φορείς, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τέταρτον, η δημιουργωντας εναλλακτικους φορεις οπου αυτο ειναι απαραιτητο η κινα παρουσιάζει την εξωτερική της πολιτική όλο και περισσότερο ως μια εναλλακτική άποψη σε σχέση με την αντιμετώπιση που βασίζεται σε αξίες για τους τωρινούς διεθνούς, διεθνείς φορείς που υποστηρίζονται από την Ευρώπη και το δυτικό κόσμο. Επομένω η Κίνα όλο και περισσότερο τονίζει τις δικές της αρχές, ιδίως την κυριαρχικότητα και την μη παρέμβαση ως βασικές αρχές για την διεθνή συνεργασία των κρατών. Εγώ θα σταθώ τώρα σε τρία μοναχα στοιχεία από τη μελέτη μας. Πρώτα απ' όλα την Κίνα με την, και τις σχέσεις της με την παγκόσμια διακυβέρνηση, δεύτερον την Κίνα και τις εδαφικές διαμάχες στο νότιο κινέζικο πέλαγος και τρίτον την Κίνα και την ευρωπαϊκή γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, στα θέματα διεθνούς διακυβέρνησης, όπως είπα προηγουμένως, η Κίνα αμφιταλαντεύεται μεταξύ του να επιβεβαιώσει από τη μια μεριά τους υπάρχοντες φορείς διεθνούς διακυβέρνησης αλλά και τον να υποστηρίξει τη μεταρρύθμισή τους και από την άλλη πλευρά δείχνει τη θέλησή της να δημιουργήσει εναλλακτικέ δομές όπου δεν μπορεί να ασκήσει πράγματι την επιρροή της στους διεθνείς φορείς. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση των φορέων διεθνού διακυβέρνηση, μπορούμε να πούμε ότι η Κίνα ικανοποιημένη με την παρουσία τη ω μόνιμου μέλου του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν ζητά περαιτέρω μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας παρά το γεγονός ότι ρητορικά υποστηρίζει την πολυπολικότητα. Η Κίνα επίσης έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και τονίζει με αυτόν τον τρόπο το ότι αποδέχεται τον ΠΟΕ ως τον κύριο πολυμερή φορέα για τη διακυβέρνηση του παγκοσμίου εμπορίου. Δεύτερο σημείο, η Κίνα έχει ασκήσει πίεση σε ορισμένου πολυμερεί φορεί για να μεταρρυθμιστούν, όπως παραγωγός χάρη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου η Κίνα ζήτησε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της και όταν δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το πακέτο μεταρρυθμίσεων του 2010, η Κίνα έχει καταγάγει μια σχετική επιτυχία μεταρρύθμισης του Δούνου του. Τρίτη διάσταση είναι το να ξεπεράσει, να παρακάμψει την παγκόσμια διακυβέρνηση. Η δημιουργία της Τράπεζες Επενδύσεων των BRICS και της ε, ε, Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων σε Υποδομές δείχνει το ότι είναι αποφασισμένο το Πεκίνο να ξεφύγει, να παρακάμψει τους ε, τωρινούς φορείς οικονομικής διακυβέρνησης που υποστηρίζουν τη λεγόμενη συνένεση της Washington και να τονίσει τη δική της επιρροή. Η δημιουργία της AIIB, της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων, επενδύσεων, επενδύσεων, δείχνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν για πρώτη φορά ένα φορέα, ο οποίος μπορεί να πάρει παγκόσμια υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες δεν έδειξαν να ικανοποιούνται από κάτι τέτοιο. Αν λάβω υπόψη επίσης τις διαμάχες με τις άλλες χώρες στο νότιο κινέζικο πέλαγος, εδώ βλέπουμε ένα χώρο ναυτικής επέκτασης της Κίνας. Η Κίνα διεκδικεί ή επαναδιεκδικεί την κυριαρχικότητα για ορισμένα νησιά και θαλάσσιες ζώνες που επίσης διεκδικούν άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Πέραν όμως αυτών των εδαφικών διαμαχών στο νότιο κινέζικο πέλαγος είναι σαφές ότι αναδύεται ως ναυτική δύναμη η Κίνα πέραν του δρόμου του μεταξύ στη θάλασσα τον 21ο αιώνα οι προσπάθειες της Κίνας καθοδηγούνται από την ανάγκη να βρουν νέους, πρώτους, νέους βασικούς πόρους και πρώτες ύλες και θαλάσσιες οδούς, αλλά επίσης και την διεκδίκηση ασφάλειας στην γειτονιά της. Υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτή την προβληματική. Θέλω να τονίσω το γεγονός ότι η Κίνα δεν έχει δεχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια παραπομπής στο, στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, UNCLOS, και δεν έχει δεχτεί και τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον νόμο της θάλασσας παρά τις προσπάθειες ε, των Φιλιππινών να υπάρξει μια διαιτητική διαδικασία βάσει του παρατήματος 7 του, της UNCLOS και έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό στην εκθέση μας. Τέλος, η Κίνα εμπλέκεται και στην, εσωτε... στην ανατολική γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κίνα όλο και περισσότερο είναι σημαντικός παίκτη στην γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το εμπόριο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επιλογές πολιτικών ασφαλείας. Η κρίση στην Ουκρανία έχει θέσει την Κίνα σε κάπως δύσκολη θέση, σε μια ευαίσθητη θέση σε ό,τι αφορά το σεβασμό για τις λεγόμενες πέντε αρχές της ειρηνικής συμβίωσης που υποστηρίζει η Κίνα επισήμως στις δηλώσεις της, στο Συμβουλίο Ασφαλείας κτλ. Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια ουδέτερη και εξισορροπημένη θέση. Αλλά έμεσα έχει δείξει κατανόηση για τη ρωσική θέση. Και η άποψη της Κίνας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ κοντά στην ρωσική επίσημη άποψη, ενώ η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για τα θέματα της Ουκρανίας δεν είναι ικανοποιητική. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ο παράγον των ρωσοκινέζικων σχέσεων. Η υποστήριξη της Ρωσίας είναι πολύ σημαντική για την, ε, Ρωσία, είναι σημαντική για την ε, Κίνα, <clears throat> γιατί αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παροχή φυσικού αερίου, εξελιγμένα όπλα, αυξημένο εμπόριο και καλύτερη και ισχυρότερη γεωπολιτική υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν οι ίδιες αξίες της πολυπολικότητας και της μη παρέμβασης για στις δύο χώρες, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την πρόθεση των συμφερόντων τους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε φορείς όπως είναι το G20, η BRICS κτλ σε περιφερειακό επίπεδο, αν εξαιρέσουμε την Κεντρική Ασία, δεν έχουν διαμάχες, δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τους, κάτι το οποίο βοηθά αυτές τις πρωτοβουλίες. Τέλος, η Κίνα έχει αναλάβει την πρωτοβουλία του δρόμου του μεταξιού στην Κεντρική Ασία, που θέλει να θέσει την Κεντρική Ασία ως ένα νέο διάβλο μεταξύ από Ανατολής και της Ευρώπης. Επομένως βλέπουμε μια μορφή επαναπροσανατολισμού από μια προσέγγιση μεγάλης δύναμης και μόνο σε μια δημιουργία συνεργασίας με άλλες χώρες της Ασίας, δημιουργία εναλλακτικών δρόμων εμπορίου που θα μπορέσει να αναπτύξει και τις δυτικές επαρχίες της Κίνας και καλύτερη εξασφάλιση των ενεργειακών προσόδων της Κίνας στην Κεντρική Ασία. Όλα αυτά λοιπόν είναι βασικά στοιχεία των πορισμάτων μας στην μελέτη μας και με μεγάλη χαρά θα συζητήσω σε σχέση με τις κύριες συστάσεις μας σε επίπεδο πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση ασφαλώς, όχι μόνο σήμερα. Έχουμε αρκετούς ε, σκιώδεις εδώ νομίζω. Κύριο Αντώνιο Λόπες Ιστιούρες. Σας βλέπω, τον βλέπω μάλλον στον κατάλογο των ομιλητών ως σκιώδη. Ιδάλλως ο κύριος Μποστινάρου που είναι μόνος που έχει στήσει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση και ξεκινώ λέγοντας ότι όντως ότι έχει ε, αναγνωρίσει τις, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο ευθύρες της η Κίνα και έχει τιμήσει δεσμεύσει της ή έχει τεθεί ενώπιον της πραγματικότητας με όρους realpolitik και όπου και οι δύο πλευρές πρέπει να προσδορίσουν από κοινού τις στρατηγικές τους σχέσεις. Υπάρχουν ζητήματα που ανέφεραν ήδη κάποιοι ομιλητές εγώ θα επαναλάβω τη σημασία της σχέσης αυτής με τον προσδιορισμό των οικονομικών τιμών, όπου η Κίνα συνεργάζεται με την Ευρώπη προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία και στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον επίσης. Όταν στην Κοπενχάγη, χωρίς να υπάρχει συνεργασία με την Κίνα αποτύχαμε ως Ευρώπη να διαδραματίσουμε ένα πιο ορατό ρόλο και από την άλλη βλέποντας ότι με καλύτερη συνεργασία με την Κίνα μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες ε, συμφωνίες στο Παρίσι για την παγκοσμία διάσκεψη. Πρέπει λοιπόν και οι δύο πλευρές να κάτσουν μαζί, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν ποια είναι, ποιοι είναι οι στρατηγική στοχή. οι κοινοί στρατηγικοί στόχοι. Ένα άλλο σημαντικό θέμα η Κίνα προχωρεί πολύ γρήγορα σε ορισμένους τομείς και εκφράζει ξεκάθαρα τις θέσεις της. Θα κλείσω αμέσως, Πρόεδρε. Παρακαλώ λοιπόν και καλό τους πάντες να κοιτάξουν την Κίνα με μια πρακτική, ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να κρίνει την άλλη με τα δικά της κριτήρια. Θα ήταν ε, ε το να κρίνουμε εμεί την Κίνα με τα δικά μας κριτήρια. Αλλά από την άλλη, όπως κάνουν ορισμένοι διμερό, Γερμανία, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο παραδείγματι που έχουν τεράστιου συμφέροντο διμερεί συμφωνίες με την Κίνα και προχωρούν, θα ήταν καλό να ξεκινούμε διαπραγματεύσεις για τις διμερείς συμφωνίες επενδύσεων με βάση κανόνες κοινούς για τα 28 κρατη να μην υπάρχουν κανόνες που ισχύουν για ολίγους μόνο. Εδώ δεν θα συμφωνήσω ότι ε, έχει διαιρετικό ρόλο ή διχαστικό ρόλο η Κίνα στην Ανατολική Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι οι διμερείς συμφωνίες όταν είναι προς το συμφέρον ορισμένων κρατών μελών είναι καλές. Χρειάζονται λοιπόν κανόνε και για τις 28 όταν κάνουμε συμφωνίε. έστω και διμερεί με την Κίνα. Ευχαριστώ, Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο για τις οποίες είναι καλό να έχουμε πραγματιστική ή ρεαλιστική προσέγγιση, να μην κοιτούμε μόνο δηλαδή ορισμένους όρους. Θα ήθελα λοιπόν να φερθώ σε μία πτυχή εδώ, που δεν ακούγεται πολύ. Και αυτή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί η πολιτική να μην είναι η πιο σημαντική πτυχή λοιπόν στη ζωή μας. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Κίνα. Ξέρουμε ότι μεταξύ Πεκίνου και Αγίας Έδρας δεν υπάρχουν σοβαρές διπλωματικές σχέσεις, δεν υπάρχει επαρκής αναγνώριση των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Κίνα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους ομιλητές μας, τους καθηγητές εδώ, τι είδους προοπτικές μπορούν να διαγνώσουν και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν μπορούμε να διαδραματίσουμε, σε, διαδραματίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Και θα συμφωνήσω σε κάτι που ακούσαμε από τον προλαλήσαντα, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε πραγματιστική προσέγγιση, αλλά θα πω ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να υλοποιούν, να χαίρουν πλήρως των δικαιωμάτων τους. Ναι, μπορεί κάποτε να πρέπει να ακούγεται και ο ψόγος. Όταν όμως οι συνθήκες διαβίωσης είναι κακές, πρέπει και σε αυτό να στραφούμε. Για να το αλλάξουμε. Πραγματισμό σημαίνει να μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι δεν πάει καλά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών, διδάλλως θα προλάβουμε, γιατί πρέπει να αφήσουμε αρκετό χρόνο στους ομιλητές μας. κύριος Πρατ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε μόνο η μορφή των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, αλλά και άλλες μορφές συνεργασίας των 16 συνενός επί παραδείγματι, εκ, το, εκ της οποίας βλέπουμε ότι ορισμένες από τις 16 χώρες ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες από τα Δυτικά Βαλκάνια και ταυτόχρονα υποστηρίζουμε όλοι μια ενιαία, μια ισχυρή εξωτερική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πώς μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το ειδικό φόρματ συνεργασίας των 16 συνενός. Και εν γέννη πώς κρίνετε την κατάσταση της διπλωματικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε κάπου ελλείψεις, ανεπάρκειες, κινδύνους, εάν συνεχίσουμε τη συνεργασία σε τέτοιου ίδιου φόρματ στην αυτήν αυτή περίοδο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Ευχαριστώ. Καστάλτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισέλθουμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά δύο πτυχές που είναι αρκετά προβληματικές. Η πρώτη αφορά τα πυρηνικά θέματα. Προσφάτως είχαμε τις ε, δηλώσεις του φυσικού Χέγγ ο οποίος ε, είπε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας είναι μια τρελή κούρσα ε, για να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες η Κίνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά τη διακοπή των προγραμμάτων που είχαν γίνει από το ατύχημα της Φουκουσίμα, γίνεται λόγος για ε, παραγωγή 200 γιγαβάτ ε, πριν το τέλος του 2020, κάτι το οποίο φαίνεται ότι από επιστημονική σκοπιά ε, δεν είναι δυνατόν και αυτό δηλώνει και ο Κινέζος εμπειρογνώματος. Και αυτό φυσικά θα έχει και συνέπειες για την ασφάλεια. Από τα όσα είπε ο Κινέζος φυσικός δεν θα υπάρχει δυνατότητα με τόσο γρήγορη ανάπτυξη να υπάρχουν κατάλληλα επίπεδα ασφαλείας και ξέρουμε ότι συμμετέχουν στην κατασκευή αυτού του πυρηνικού αντιδραστήρα και αρκετές ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τις νήσους Πέκλη, γιατί εκεί ε, τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια σημαντική στρατιωτική παρουσία και αύξηση τη στρατιωτική παρουσίας και ε, ένα νέο διάδρομο προσγείωσης ο οποίος ε, από ό,τι φαίνεται ε, θα μπορούσε να φιλοξενήσει ε, λόγω του μήκους του ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις, κάτι το οποίο έχει βάλει σε σκέψεις τους γείτονες από την περιοχή και φυσικά είχαμε και αρκετά αποφασιστικές δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης Ομπάμα. Τι κίνδυνος υπάρχει να υπάρξει κλιμάκωση σε σύντομο χρονικό διάστημα στο θέατρο επιχειρήσεων εκεί και επίσης ε, θα ήθελα να σταθώ και στο δράμα του λαού του Θιβέτ, διότι ε, πρόσφατα είχαμε το 140 ε, θύμα, το οποίο θυσιάστηκε για το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν χιλιά, δεκάδες χιλιάδες ε, πρόσφυγες ε, λόγω του σεισμού στο Νεπάλ και θα ήθελα να ξέρω τι πρωτοβουλίες ανέλαβε ε, η κινέζικη κυβέρνηση επί του ζητήματος. Ήσασταν πιο σύντομος από την πρώτη φορά. Ο Γιολάινον, παρακαλώ να μην μιλήσετε πολύ. Ω σκιώδη για του σοσιαλιστέ, <clears throat> είπατε κύριε Πίκε ότι οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει δεν οδηγούν κατευθείαν σε πολιτικέ μεταρρυθμίσει. Το ερώτημά μου είναι πώς προχωράει η κοινωνία των πολιτών στην Κίνα, η ΜΚΟ και τα λοιπά. Έχετε λοιπόν την ελπίδα ότι γίνεται κάτι και η καταστολή η οποία εξασ... εξακολουθεί να υπάρχει θα επικρατήσει ή θα ξεπεραστεί. Επίσης είπατε ότι υπάρχουν αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μεταφέρονται στην Κίνα. Μήπως και η Κίνα θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι διαφορετικό. Αναφερθήκατε σε χώρες όπως αυτές της Κεντρικής Ασίας και της γειτονιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, τον καθηγητή κύριο Βάλτερς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έχει εκπλαγεί με τις πρωτοβουλίες της ε, Κίνας, την αναπτυξιακή τράπεζα της ε, Ασίας, παραδείγματος χάρη. Επίσης, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής, η άποψή σας για το δρόμο του μεταξύ. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα κάποιος, <clears throat> κάποια ευρωπαϊκή αντίδραση. Είσαστε σκεπτικιστή σε σχέση με αυτά ή όχι, κύριε Βάουτες. Μίκε, θέλω να υποστηρίξω και τον τελευταίο ομιλητή τον καιρό της Σοβιετικής ε, Ένωσης λέγανε πότε θα γίνει η Αρμενία, θα φτάσει η Αρμενία το επίπεδο ζωής της ε, Ελβετίας και η απάντηση ήταν όταν υιοθετεί στο σοσιαλισμό η Ελβετία. <clears throat> Τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε αν ποτέ η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα φτάσει το ρυθμό της ε, Κίνας. Αυτό θα γίνει όταν εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές στην Κίνα. Αντί να δώσουμε τις δικές μας αξίες στην Κίνα, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κίνα να φέρει εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη να μας βοηθήσει να ξαναστάσουμε στα πόδια την κλειδονιζόμενη οικονομία μας και πώς οι ιδέες αυτές της Κίνας να εφαρμοστούν μέσα στην Ευρώπη και να ξεπεράσουμε την οικονομική καταστροφή που έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί θέλουν να σκεφτούν κάτι τέτοιο πρέπει να θυμηθούν ότι το ΑΕΠ της Ευρώπης στο κατακεφάλι είναι πολύ, πολλαπλάσιο αυτό της Κίνας. Δεν πρέπει να μιλήσετε για αριθμούς ανάπτυξης. Πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι και τα σημεία εκκίνησης των δύο οικονομιών. Και σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κινέζικων αξιών, καλή τύχη και καλά κρασιά. Ο κύριος Ουχελή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αντιπροσωπώ τον ε, εκπρόσωπο της ομάδας μας για την... Ε, είμαι μέλος της Επιτροπής, εν της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Αντιπροσωπείας της Κίνας. Και έχω σταθεί ε, αρμόδιος στην Ουγγρική κυβέρνηση για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις Ουγγρικ... συνοουγγρικές σχέσεις. Βλέπω λοιπόν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Βλέπω ότι έχει πραγματικά νόημα το να έχουμε μια καλή σχέση με τους ε, Κινέζους. Την τελευταία μισή ώρα ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για την Κίνα. Αλλά έχουμε αναλύσει και την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς εμείς στεκόμαστε αυτή τη στιγμή ενώπιον της πραγματικότητας στην Κίνα και πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μελλοντική εξέλιξη της Κίνας. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα προς τον εισηγητή μας. κατά πόσο τα στρατηγικά μας σχέδια έχουν λάβει υπόψη και τις ε, συνέπειες που προκύπτουν από μια κοινή αντιμετώπιση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ομφαλοσκοπεί. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί ζηλεύουν τους Ρουμάνους και τους Ούγγρους όταν κάνουν ειδικέ ε, συμφωνίες με το Πεκίνο, αλλά δεν γίνεται το αντίθετο. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες και αυτές θα πρέπει να υποστηρίξουν, πρέπει μόνο οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δικές τους συμφωνίες και όχι οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν όλοι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την αναδυόμενη Κίνα και να μην θέσουμε τον εαυτό μας σε μειονεκτικό έδαφος. Ευχαριστώ. Please. <clears throat> Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, ιδιαίτερα στις ε, τοπικές κυβερνήσεις, ποιο είναι το επίπεδο της διαφθοράς Δεύτερη ερώτηση, γιατί επιστρέφω από τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Απαγόρευσης των Πυρηνικών. Ποια είναι η στάση της Κίνας σε σχέση με το Ιράν και ποιες είναι οι τάσεις σε σχέση με, τον πυρηνικό, με τους πυρηνικούς εξοπλισμούς στη Μέση Ανατολή. Πρόεδρος, οι πυρογνωμόνες λοιπόν τώρα, από δύο λεπτά ο καθένας, λυπούμε, ξέρω ότι δεν είναι σοβαρό να σας δίνω τόσο λίγο χρόνο, κακός προγραμματισμός από πλευράς μας. Με αντίστροφη σειρά τώρα, καθηγητής Waters. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, δεν είναι πολύ χρόνο στα δύο λεπτά, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα. Ο μέσος χρόνος ομιλίας για, το, για τους ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια είναι το ένα λεπτό να ξέρετε. Α, τιμή μου τότε. Λοιπόν, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Κίνα. Βεβαίω ε, είναι πολύ γνωστό το ζήτημα ε, στι σχέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κίνας, με ό,τι μορφή και να έχουν πάρει. Είναι μακροσκελής και διαρκούν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η Κίνα μαζί με τη Ρωσία θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτή την προσέγγιση, την αξιακή και προσπαθούν να ορίσουν μια διαφορετική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα, ακανθώδες και πολύ σημαντικό θέμα πολιτικής που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ποιος είναι ο αντίκτυπος δηλαδή στο, του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα και όπως εμείς ε, συστήνουμε θα ήταν καλό ενδεχομένω να ενθαρρύνουμε και την ε, ένταξη της Κίνας σε ένα άλλο ε, διεθνή οργανισμό ή φόρουμ ή άλλων ε, φορέα ε, βάσει του κράτους δικαίου που είναι από τους τρεις βασικούς πυλώνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το, και της διεθνής της σχέσης και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο σημείο εκκίνησης για να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε το πεδίο της εταιρικής συνεργασίας. Τώρα για τα όσα αναφέρεται για το 16 είναι 1, Πράγματι είναι μια ενδιαφέρουσα δυναμική που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Κίνας και της ε, περιφέρειας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ ενδιαφέρον ως ε, δίκτυο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η γραμματεία αυτού του 16 συν 1 εδρεύει στο Πεκίνο. Είναι και μια κινέζικη πρωτοβουλία δηλαδή και πράγματι υπάρχει μια ασυμμετρία σε αυτή τη σχέση. Όμως είναι σημαντική προσπάθεια και να αναφέρουμε και τις πρόσφατες τρεις γραμμές του Βελγραδίου, όπου οι εταίροι ανέφεραν ότι υπάρχει ε, η ιδέα της αμοιβαίας ωφέλειας, η συνεργασία win-win, αλλά και υιοθετούν ότι όλα αυτά συνάδουν και με την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, που είναι σημαντικός παράγοντας. Τέλος, η πρωτοβουλία της Κίνας για την ε, θέσπιση μιας νέας ασιατικής περιφερειακής τράπεζας είναι ένας από τους ε, παράγοντες που προσπάθησα να υπογραμμίζω ως ε, ένα εναλλακτικό διάβημα της ε, Κίνας για την διαμόρφωση άλλων δομών μέσω των οποίων μπορεί να επηρεάσει την μεταρρύθμιση των δομών Bretton Woods. Είναι ένα καινοτόμο στοιχείο. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, ε, προσυπογράψει, 40 τον αριθμό και θα ήταν ε, θετικό να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τη θέση μας, αλλά όχι να κλείσουμε την πόρτα σε αυτή την πρωτοβουλία. Μία μορφή επικοδομητικής συμμετοχής λοιπόν. Όχι βεβαίως το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, αλλά ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Νόμιζα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα τα πω λίγο διαφορετικά. Είναι αλήθεια ότι ε, έχουν ξεκινήσει οι σχέσεις από το 1996 στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Από ό,τι διαπίστωσα εγώ όμως, η Κίνα αλλάζει μόνο όταν συμφωνεί και όταν συνειδητοποιεί ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Επομένως, ακόμα και αν πιεστεί, δεν θα είναι αποτελεσματικό. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν ήδη συνειδητοποιήσει οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια. Το να ασκηθούν πιέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα μπορεί τελικά να έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούν. Καλό είναι να υπάρχει ένας διάλογος και ο διάλογος να συνεχιστεί μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης συμφωνώ ότι από τότε που Ζη Σιγκίνγκ ε, ανέλαβε την εξουσία, αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κίνα είναι το κράτος δικαίου και προσπαθούν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση η κοινωνία των πολιτών. Αλλά το θέμα είναι τι θα πετύχουν. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά την ερώτηση του Γιώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί συνεχώ να αλλάξει την Κίνα. Το κατά πόσον όμω η Κίνα θα θέλει να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, νομίζω ότι η Κίνα ε, είναι απασχολημένη με το δικό τη ε, το θεματολόγιο και ακόμα δεν έχει καμία επιθυμία να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η εξωτερική πολιτική της Κίνας ουσιαστικά είναι προέκταση της εσωτερικής της πολιτικής, επομένως ό,τι και να κάνει η Κίνα γίνεται γιατί συνειδητοποιεί ότι πρέπει να το κάνει. Με άλλα λόγια, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την κατάσταση της Κίνας, ε, την πολιτική της Κίνας, τα δικά της τα προβλήματα και να αντιληφθούμε ε, ότι η εξωτερική της πολιτικής έχει σχέση με όλα αυτά και με τη σχέση της Ευρωπαϊκή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτό θα σταματήσω. Κύριο Πίκη. Ναι. Να μιλήσω κι εγώ για τα δυο λεπτά μου αυτά της δόξας που μου παρέχεται. Καταρχάς, η προσέγγιση στη σχέση με τις Κίνες και το κατά πόσο θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτεί τι θέλει να επιτύχει στη σχέση της με την Κίνα και σε συνεργασία με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από... Μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Κίνα, ιδίω από την κυβέρνηση, διότι θεωρείται ότι είναι κατακαιρματισμένη και δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέλει και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον αν δεν υπάρχει δημοκρατία στην Κίνα πρώτα θα πρέπει να δούμε τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας για το μέλλον και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Το κράτος δικαίου αναφέρθηκε επανειλημμένος και αυτό είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Ε, είναι ένα θέμα υπαρκτό Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε Κινέζοι όμω, ε, δικηγόροι οι οποίοι ε, ζουν ακριβώς από το κράτο δικαίου στην Κίνα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως νομίζουμε. Επίσης υπάρχει μια ε, δημοκρατία η οποία κατευθύνεται και περιορίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και μέσω αυτής της κατεύθυνση και αυτών των περιορισμών υπάρχουν ε, πολλές φορές πολύ σοβαρές ε, συνέπειες για την πολιτική, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, σε πολλά τμήματα της Κίνας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η κινέζικη κυβέρνηση και ε, ο Τσι προσπαθεί να διαμορφώσει την Κίνα ε, και όχι περισσότερο να την κυβερνήσει. Προσπαθεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Δημιουργεί μια νέα κοινωνία η οποία θα συμμορφούνται περισσότερο στην εικόνα που έχει ο ίδιος για το πώς θα πρέπει να είναι η κινέζικη κοινωνία και νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό προκειμένου να δούμε πώ θα είναι η Κίνα στο μέλλον. Μια κοινωνία η οποία δεν θα είναι απλώς ε, ένα σύνολο ατόμων ή προσωπικών συμφερόντων, αλλά θα γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο το οποίο ε, κυβερνάται από ένα σύνολο κοινών κανόνων και στόχων και στην πραγματικότητα αυτό είναι το σκεπτικό ε, το οποίο θα τους ε, κατευθύνει, το οποίο είναι διαμέτρου αντίθετο από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι δυτικές χώρες της κοινωνίας τους. Ευχαριστώ για σε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και ως εισηγητής ε, για τα θέματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συμμετέχοντες για την ε, πολύ καλή συμβολή τους. Ανέφερε και ο κύριος Επίκε ε, το πρόσωπο της Κίνας και ποιο πρόσωπο εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο. Πολλές φορές αναφέρθηκε το κράτος δικαίου, εξαιρετικά σημαντικό να το εξετάσουμε, όμως βέβαια θα πρέπει, όπως έκανε και ο κύριος Πίκε, να δούμε τι ακριβώς εννοούμε κράτος δικαίου. Δεν είναι μόνο ο νόμος. Αν θέλουμε να πούμε στα σοβαρά τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο σοβαρά με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και κλείνοντα Πρόεδρε, που ανέφερε και ο συνάδελφο Οστινάρου και άλλοι, ότι εάν θέλουμε, είναι σημαντική για μα αυτή η εταιρική σχέση, θα πρέπει να βρούμε καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι να το εξετάσουμε κατακαιρματισμένα σε κάθε κράτος μέλος, όπως έγινε με την Επενδυτική Τράπεζα στην Ασία όπου υπήρξε και πάλι έλλειψη συντονισμού. Να μιλούμε λοιπόν με μία ενιαία φωνή, με καλύτερο συντονισμό για τα σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος της διεθνής μας σχέσης με την Κίνα, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση και μας δίνει και πολλές ε, προοπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλλορ. Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ε, συμμετοχή της Κίνας στους διεθνείς φορείς με τον τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με την Κίνα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονές μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση σε βάθος χρόνου και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Παρά την πίεση χρόνου και σας ζητώ συγγνώμη για την τελευταία αυτή πίεση χρόνου. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, της ψηφοφορίες, έκθεση ΣΑΚΕ καταρχήν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία. Θέλεις Μαρίτσια να πεις κάτι σχετικά? Όχι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίες. 26 με 32 απορρίπτεται. 44. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται 37-27. Τροπολογία 46. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την διαπλειοψηφία. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 49. Ψήφι υπέρ. Υπέρ 49. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά Α, εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. φοφοριες ψηφοφορίες. 36-30 γίνεται δεκτή. 54 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρασης ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35-29. Περνάμε στην τροπολογία 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ίδια πλειοψηφία λέει ο πρόεδρος. Λυπάμαι, δεν χρειάζεται έλεγχος. Γίνεται, έγινε η ψηφοφορία, ψηφοφορια ψηφοφορίας. 34-30 έγινε δεκτή παρόλα αυτά. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. 98 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. 29-19 γίνεται δεκτή. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος βεβαίως. Αφού οι φιλελεύθεροι άλλαξαν γνώμη, πέρας 31-35 απορρίπτεται, μάλιστα. Δεν τους, ε, τους υπερεκτίμησα τους φιλελεύθερους, λέει ο πρόεδρος. 104. Ναι, έχει γίνει δεκτή κάποια από τις προηγούμενες τροπολογίες που αναφέρετε εδώ. Εντάξει, δεν ψηφίζουμε. Αυτή είναι 106. Υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. 37-28 εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γίνεται δεκτή, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Δεκτή, δεκτή, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 110 υπέρ. Υπέρ, κατά, Τι, τι ψηφίζετε, υπέρ ή κατά τώρα. Εγκρίνεται. 111 Χέγγελ υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 111. Henkel 111. Πέρας. 28 με 36 απορρίπτεται. 100 ήταν Χένκελ αυτή. Ναι. 112 υπέρ. <clears throat> Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 113 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 117 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Πάμε. Συμβαστική 16 η ηλεκτρονική ψηφοφορία ελέγχου. Πέρας εγκρίνεται 37-25. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 129. Υπέρ. Πάλι. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι σαφές. 130-131. Υπέρ. Είναι ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 133. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135, 36 και 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες της κυρίας Σάκε 146 μέχρι 152, όλες μαζί. 146 με, ναι, παρακαλώ. Όχι. ...46, 47, 48 μέχρι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 κατά αποχές εγκρίνεται, 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 18 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 163 υπέρ κατά α, έλεγχος για την 163. Πέρας ψηφοφορίας. 28-36 απορρίπτεται, 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, 167 υπέρ, κατά Ορίστε. Ένα μπλοκ με τις ε, τροπολογίες Βάιντενχόλτσερ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, λέει ο πρόεδρος. 1.64 μέχρι 176. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Αποχές. Έλεγχος καλά. οι FTD έχουν ένα πλεονάζοντα. Ψηφίζει ένας παραπάνω. Προσπαθήσατε κύριε Καστάντο, αλλά δεν έπιασε. Πέρα της 35 με 28 εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, «20 και 21 μαζί, μπορούμε, ναι. Υπέρ 20 21. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 μέχρι 27 μαζί. Μπορούμε. 23 έως 27 από κοινού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτή ήταν 31. Ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας της 25 με 31 απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται μάλλον, λέει ο πρόεδρος. 35. ποιο είναι υπέρ. Επαναλαμβάνει η ψηφοφορία ο πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Ναι, ναι, απορρίφθηκε. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή, τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή, πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτή, έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή, εφτά υπέρ κατά αποχές δεκτή, οχτώ υπέρ κατά αποχές δεκτή, εννέα υπέρ. Καλά έλεγχος μέσα ναι, στην οκτώ. Πέρας ψηφοφορίας. 33-28 εγκρίνεται πράγματι. Το έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 33 υπέρ. 6 κατά. Αρκετές οι αποχές 24. Εγκρίνεται. 28. Äh, der Kollege Chip, haben Sie noch etwas zu sagen? Έχετε τίποτα άλλο να πείτε σε αυτό. Για το θέμα σας κύριε Ξούπ, έχετε τίποτα να πείτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη διευκρίνηση ή επεξήγηση. Θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην τροπολογία 25 στην αιτιολογική σκέψη H έχω μια προφορική τροπολογία και είναι προφορική ο πρόεδρος ο διακόπτη Κοιτάξτε τότε όταν έρθει η ώρα του να το εξηγήσετε. 28 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 34 κατά, Απερίφθη συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Δεν είναι πολύ σαφές. 33 πάλι. Κατά. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Έρας. 28 υπέρ, 29 κατά, απερίφθη. Σωστά έλεγα εγώ. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 42 τμήματα, πρώτο τμήμα παρακαλώ, κατά αποχές απερίφθη, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, και πάμε στην 48 ε, υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 6 συμβαστική υπέρ. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έκανε ένα λάθος. Έπρεπε να είχαμε ψηφίσει 47. Αλλά το κάνουμε και τώρα μένα. Υπέρ λοιπόν τη 47. Κατά. Αποχή συγκρίνεται. Και πάμε στην 54 τώρα, δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Δεύτερο υπέρ, κατά, υπέρ πάλι, υπέρ στο δεύτερο τμήμα της 54. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές Επαληθεύουμε. Πέρα της ψηφοφορίες. 26 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 57 υπέρ, κατά, επαληθεύμα. Πέρας. 26 υπέρ 32 κατά. Απερίφθη. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 66 δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 68 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 69 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 70 υπέρ κατά επαληθεύουμε. Πέρα τις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Εδώ το 69 το οποίο περίφθη είχε την ωραία ιδέα ότι κάποιος ε, που χτυπάει τη γυναίκα του μπορεί να το, αρνηθεί στο πλαίσιο της, ε, των θεμάτων για τη δημοκρατία. Πάμε στη συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ 11. Την 11 θέλετε να επελθεύσουμε. Antrag ist Gott sei Dank angenommen, äh, ist angenommen worden. Dann grünete. Γιατί να μην μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκευτικέ μειονότητε σε περιπτώσει όπου διώκονται χριστιανοί, δεν το καταλαβαίνω. Τώρα πάμε στην 81. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 82 δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές Απερίφθη. 15 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 101 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε. Πέρα της ψηφορίες. Μάλιστα. 17, συμβαστική 17, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Όχι 5. 5 στην 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 λέει ο πρόεδρος, συμβαστική πρέπει να εννοεί, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 12, τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται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 Η 25 ήταν με την προφορική τροπολογία. Ναι, όπως την έχουμε στο κατάλογο μας. Η 25 έχει με την προφορική της τροπολογία εγκριθεί. Είναι στο κατάλογο. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Υπαριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Das war 11, 53 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά, μία αποχή. Και συγχαρητήρια, κύριε Ισηγητά, και βέβαια στην κυρία Σάκη για την προηγούμενη έκθεση. Και άρα λίγη η συνεδρίασή μας. Καλό σας βράδυ.